Αρχίζουμε τη σημερινή μας συνεδρίαση με τις ψηφοφορίες. Ελπίζω να έχετε φέρει όλοι μαζί σας ε, την κάρτα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Για να ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία της προφορικής ερώτησης με θέμα τη διάσταση των φύλων ε, την εμπορία ανθρώπων. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σημείο 12. Χειραφέτηση των κοριτσιών μέσω της παιδείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 69. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές θα κάνουμε ένα ηλεκτρονικό έλεγχο άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 69 τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται 11 ψήφι υπέρ 13 κατά 70 ποιος είναι υπέρ τροπολογία 70 κατά Αποχές εγκρίνεται. 71. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 72. Ποιος είναι υπέρ. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Πρώτη 17 της Επιτροπής Πολιτισμού. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 72. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 72 άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται τροπολογία 73 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 76 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 77. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 83 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 81 τώρα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 85 με προφορική τροποποίηση της συγκεντρές ποιος είναι υπέρ κατά εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 89 παρακαλώ άρχεται ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται Τροπολογία 90. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 91 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 106. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. 22 της Επιτροπής Πολιτισμού. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ κατά άποχες ηλεκτρονικός έλεγχος για την 114 παρακαλώ άρχεται ψηφοφορία τέλος απορρίπτεται με μία ψηφοδιαφορά. συμβαστική τροπολογία 10 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 11 της Επιτροπής Πολιτισμού. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 120. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 122 σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της 122. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 125. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 12. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 της Επιτροπής Πολιτισμού. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8 της Επιτροπής Πολιτισμού. Υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 8 της Επιτροπής Πολιτισμού έρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 132 ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 142 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα της 142 144 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 145 με προφορική του απολογία της ηγετρίας που έχει περιληφθεί στο κείμενο ποιος είναι υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 145 άρχεται η ψηφοφορία Τέλος ψηφοφορίας Απορρίπτεται. 146. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 175 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 175. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται, αλλά παρακαλώ κάντε τον κόπο να σηκώνετε τα χέρια σας γιατί δεν είμαι και μάντης. 155 και 156 πανομοιότυπες. Ε, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις 155 και 156. Τέλος ψηφοφορίας. Ε, ήρθατε στην κατάλληλη στιγμή κύριε Ταραμπέλα. Απορρίπτεται. Τέσσερα της Επιτροπής Πολιτισμού ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 158 ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 159 υπέρ. Εκατόν πενήντα εννέα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εκατόν εξήντα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εννέα της Επιτροπής Πολιτισμού υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκατόν εξήντα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 164 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 165 έχει αποσυρθεί 166 τώρα ποιος είναι υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 167 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 167 υπέρ. Mm. 163. 163. Με προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δύο της Επιτροπής Πολιτισμού υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 169 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 171 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 174 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 176 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 176 άρχεται η ψηφοφορία τέλος εγκρίνεται Οπότε περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 18. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 180. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 181. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 182 έχει αποσυρθεί. 183 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 183 άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 185 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 186. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 187 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 188 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 189 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται και αυτό. Συμβαστική τροπολογία 19. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 194. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 194. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 195. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 196. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 197. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 198. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 199 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 200 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 200. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Ωραία. Πέρας. Απορρίπτεται. 201 ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 202 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στη συμβαστική 20 Ψηφιπέρο. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 206 ψήφι κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 ψηφιπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή τροπολογία 8 ψηφιπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 10 ψηφιπέρ, κατά αποχές ας κάνουμε επαλήθευση τροπολογία 10 ψηφιπέρ, πέρας δεκτή πέρας σε τροπολογία 11 υπέρ κατά αναποχές δεκτή τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 13 ψηφιπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 14 ψηφιπέρ κατά αποχές Ας επαληθεύσουμε τροπολογία 14, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15 ψηφιπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 16 υπέρ. Συγγνώμη. Τροπολογία 19. Τροπολογία 19 ψηφιπέρ κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική τροπολογία 2 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 3 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 22 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 24 ψηφιπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 27 ψηφι Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 23 ψηφι Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 25 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα ψηφι Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα ψηφιπέρ Κατά. Αποχές. Δεκτό. Τρίτο τμήμα ψηφιπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπερθμών 26 ψηφιπέρ Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία υπερθμών 29 ψηφιπέρ. Συγγνώμη, 28. Ψηφίζουμε επί της 28. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 29. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίτεται. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Παρθμό 31 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Προπολογία 32 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Υπερθμό 34 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Υπάρχουν 36 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό 37 υπέρ κατά αποχές δεκτό Υπερθούν 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Υπερθούν 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στη συμβαστική 4, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές δεκτό. Περνούμε 44, υπέρ. Κατά, αποχές δεκτό. Περνούμε 46, <clears throat> υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά, αποχές Ας επαληθεύσουμε επί της 48. Άρχεται ψηφοφορία. Ε, απορρίπτεται. Περιθμός 47 ψηφί υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Παριθμόν 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ κατά αποχές δεκτή 57 υπέρ κατά αποχές δεκτή 59 υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε την 59 άρχη της ψηφοφορία απερίφθη υπερθμόν 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές δεκτή 62 υπέρ κατά αποχές δεκτή 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές δεκτή 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 1 με προφορική τροπολογία του εισηγήτρια Υπέρ. κατά εποχές δεκτή οι 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή και τώρα περνάμε στην τελική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία Πέρας εγκρίθηκε με 21 ψήφους υπέρ, 9 ψήφους κατά. Συγχαρητήρια κυρία Ροδρίκης για την έκθεσή σας. Sí, Eh, Θα περάσουμε τώρα στην επόμενη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης. Η συγγήτρια είναι η κυρία Ζαμπόσκα, η οποία θέλει σύντομα να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω, αλλά θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις ηγητές, διότι το αποτέλεσμα ήταν 13 ε, συμβαστικές τροπολογίες και θεωρώ ότι είναι μεγάλη επιτυχία. Νομίζω ότι έχουμε συμπεριλάβει πάνω από 50 τροπολογίες σε αυτές τις συμβιβαστικές και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στους σκιώδεις ηγητές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ζαπόρσκα. Περνούμε στην ψηφοφορία της έκθεσης. Η 51, πρώτη τροπολογία σε δύο τμήματα, υπέρ του πρώτου κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί, αλλά χρειάζεται έλεγχος, παρακαλώ για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας του παρελθόν 51. Πέρας. Εγκρίθηκε. 15 ψήφι Η τροπολογία παρελθόν 50. Ψήφι Κατά. Αποχές. Έλεγχος και πάλι για την 50. Άρχεται η υπολήθευση. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η τροπολογία περίφημα 53 ψηφίπε Κατά. Αποχές. Δεν σας βλέπω, δεν σηκώνετε χέρια. Έλεγχος για την 53. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. 23 υπέρ. Αν βλέπω καλά. Καταπίπτει 20. Ψηφίζουμε την 54 Είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 56 Είπε. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 57 Είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 55 Είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 58 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ, κατά, απόχες. Ηλεκτρονική επαλήθευση για το πρώτο τμήμα, λέει η Πρόεδρος, συγγνώμη, το δεύτερο. 58 άρχεται η επαλήθευση. Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα το δεύτερο υπέρ, κατά, απόχες, εγκρίνεται. Η 59 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Κατά πίπτη 60. Η 7 της απασχόλησης υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Κατά πίπτη 61. Συμβιβασμός υπαριθμών 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 65 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 66 ψηφιπέ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 73 υπέρ κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Στην 73 άρχεται η ψηφοφορία. Σε θύρα Πέρας, απορρίπτεται. Δεν θα ψηφίσουμε τη 14 της Επιτροπής Απασχόλησης. Πάμε στην 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. τροπολογία 75. Σε δύο τμήματα ψήφι υπέρ του πρώτου κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέ κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει η τροπολογία 12. Τσέκ, τι, πιανού. Τι θέλετε να τσεκάρουμε. Ωραία. Έλεγχος του δευτέρου τμήματος της τροπολογίας 75 αρχίζει τώρα ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε στην 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 3 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέ. κατά εγκρίνεται. Η τροπολογία 78 καταπίπτει. 128 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτον υπέ. Α, συγγνώμη, και αυτή καταπίπτει, διότι έχει εγκριθεί η τρία της ε, Πάμε στην 71. Υπέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 4 υπέρ της Επιτροπής Απασχόλησης κατά αποχές εγκρίνεται. Τσεκ φωνές. Λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 4 της Επιτροπής Απασχόλησης. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 52 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλαχος και πάλι. Για την 52. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σε cierra la βοτασιόν. Εγκρίνεται. 84 πίπτη, Οπότε θα πάμε στα 83 ψήφι Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 3 ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση γιατί είναι 95, αρχίζει τώρα. Τέλος. Ισοψηφία, άρα απορρίφθηκε. 96 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται. Τσεκ. Για την 96 άρχεται η ψηφοφορία. έχει απορριφθεί και με μεγάλη διαφορά μάλιστα. 96. 96 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 97 υπέρ. Όχι, 98 είναι σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο είπε κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Θα ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα της 98. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρασα. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 99 είπε κατά αποχές Ζητώ συγγνώμη γιατί είναι πολύ μικρή διαφορά. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίθηκε. Η 100 είπε. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 101 είπε. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 4 είπε κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 110 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 111 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση στην 112 έρχεται ψηφοφορία Πέρας εγκρίνεται 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 114 σε δύο τμήματα τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα υπέρ Α, όχι, καταπίπτει το δεύτερο ακούω, μάλιστα. Πάμε στο συμβασμό υπαριθμό 6, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 119 τροπολογία τώρα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 122 τμήματα τμήμα πρώτον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται φόλς φωνές ότι καταπίπτει όχι, καταπίπτει εφόσον απορριφθεί το πρώτο τμήμα το οποίο εγκρίθηκε, άρα πρέπει να ψηφίσουμε το δεύτερο. και ψηφίστηκε και πέρασε. Λοιπόν, 121 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση 121 αρχίζει τώρα. Πέρασε. Εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ah, la 121 no la hemos votado. Sí, sí, sí. Sí. Η 164 δεκα... Λοιπόν, η 164 καταπίπτει διότι 120 έχει εγκριθεί. Το ίδιο ισχύει και για τη 13 της Επιτροπής Απασχόλησης. Πάμε στη 17 της Απασχόλησης, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει η επόμενη 123. Πάμε στην 124 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. η ε, πίπτη η επόμενη 9 της απασχόλησης. 125 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 126 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 127 είναι γλωσσική και δεν ψηφίζεται. 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ορίστε. 131 ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει τώρα. Πέρας. Απερίφθη. 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 136 ειπέ, κατά, αποχές εγκρίνεται, ε, καταπίπτει 10, 138 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 137, έλεγχος για την 138, αρχίζει ηλεκτρονική επαλήθευση. Απορρίπτεται. 137 επέ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 139 επέ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 140 κατά πίπτη. 142 επέ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 143 επέ Κατά αποχές εγκρίνεται 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 145 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 6 ας συγγνώμη 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η επόμενη καταπίπτει 149 επέ κατά αποχές εγκρίνεται 150 επέ κατά αποχές δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι έγινε 150 επαληθεύουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται. 151 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 158 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 158. Άρχεται η ψηφοφορία. Τερνάμος. Ρετσαθάδα. Απορρίπτεται. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικό Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 159. Άρχεται η ψηφοφορία. rechazada. Απορρίπτεται. 160 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ. Α, συγγνώμη. Καταπίπτει 161. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 163 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19 της απασχόλησης δεν το ψηφίζουμε. 168 εντάσσεται στη συμβαστική τροπολογία. Περνάμε στην 169. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δύο της Επιτροπής Απασχόλησης. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 της Επιτροπής Απασχόλησης. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις, μάλλον αναφορές, τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται.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 εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 συμβαστική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 24. Ηλεκτρονική επαλήθεση. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 25. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 καταπίπτει 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ο β της ε, απασχόληση υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία της έκθεσης. Ψηφίσατε όλοι. εγκρίνεται με 24 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 6 αποχές. Συγχαρητήρια κυρία Ζάμπορσκα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με βάση το άρθρο 56 των διαδικαστικών κανόνων, θα ήθελα να εκφράσω την γνώμη μου, που είναι γνώμη μια μειοψηφία και θα τη διαβιβάσω γραπτός το απόγευμα στη Γραμματεία. De Pasamos a la del siguiente informe Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία της εντολής για το τριμερή διάλογο για τον προϋπολογισμό του 2016. ver, continuamos, continuamos, con la, continuamos con la votación. La señora... Συνεχίζουμε. Έχουμε και άλλη ψηφοφορία. Η κυρία Ζαμπόσκα εξέφρασε την γνώμη τη που είναι γνώμη ψηφία. Έχετε δυνατότητα με βάση τον κανονισμό. Μπορεί κάλλιστα να διαβιβάσει τη γνώμη τη που είναι γνώμη μειοψηφία στη γραμματεία για να περιληφθεί. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, προβλέπεται από τον κανονισμό. Θα περάσουμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία που αφορά την εντολή στον τριμερή διάλογο για τον προπολογισμό του 2016, γνωμοδότηση ματέρα. Τροπολογία 5, ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6, ποιο είναι υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 7, υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 8, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και 4. Ποιος είναι υπέρ. Α, έχει αποσυρθεί η 4. Τελική ψηφοφορία της νομοδοτήσεως. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. 26 ψήφισαν υπέρ, 4 κατά, χωρίς αποχές. Εγκρίνεται η εντολή για τον τριμερή διάλογο, για τον προϋπολογισμό του 2016. Ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και περνάμε στην κανονική μας συνεδρία στην υπόλοιπη.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

Disculpe. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τώρα τις εργασίες μας. Επαναλαμβάνει και στα αγγλικά η Πρόεδρος. Όσοι δεν ενδιαφέρονται, παρακαλώ να περάσουν έξω. Pasamos al intercambio de puntos de vista del Περνάμε στην ανταλλαγή απόψεων ε, τη εξέσεω ε, που έχει θέμα τις γυναίκες ε, στον επιστημονικό και πανεπιστημιακό χώρο. Η κυρία Βόζενμπερκ είναι η συγγετρία και της δίνω το λόγο για να μας παρουσιάσει την έκθεσή της. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς στην αρχή να πω ότι Έχω πλήρη συνείδηση ότι αυτή η έκθεση αφορά σε όλους και σε όλες μας και αφορά και σε κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά με το δεδομένο ότι υπάρχουν ανισότητες οι οποίες κατά καιρούς καταγράφονται σε όλες εκείνες τις υπηρεσίες ερευνών και στατιστικής. Σε κάθε περίπτωση η πρώτη μου προσέγγιση, η έκθεση έχει δημοσιευθεί προσφάτως και ε, πιστεύω ότι όλοι είχατε την ευκαιρία να τη μελετήσετε, αλλά σε κάθε περίπτωση χρονοδιάγραμμα κλειστό δεν υπάρχει, δεν μας πιέζει εξαιρετικά ο χρόνος. Ε, μπορούμε και προϊόντος του χρόνου, άλλωστε μέχρι τις 22 Ιουνίου έχουμε ε, το χρονοδιάγραμμα για τις τροπολογίες. Η έκθεση έχει χωριστεί σε επιμέρους κατηγορίες για να μπορεί να γίνει αντιληπτό από τον καθένα ε, ο τομέας στον οποίο θέλει να παρέμβει, θέλει να σχολιάσει, ούτως ώστε η έκθεσή μας να, εκφράζει ε, κατά το δυνατόν την πλειονότητα των απόψεων που έχουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Ε, η πρώτη κατηγορία αφορά πραγματικά στην ισότητα των φύλων, στην ακαδημαϊκή σταδιοδρομία και την έρευνα. Ε, παρατηρούμε ότι ενώ υπάρχουν τομείς όπου οι γυναίκες πραγματικά έχει, τους έχει δοθεί η ευκαιρία να κάνουν θαύματα, υπάρχουν άλλοι τομείς όπου είτε υποεκπροσωπούνται είτε εμποδίζονται ε, χωρίς δική τους θέληση να μπορέσουν να εκφραστούν σε ανώτατο επίπεδο ε, με βάση τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Επομένως αυτό προσκρούει άμεσα και κέρια στην αρχή της ισότητας ιδιαίτερα στην ακαδημαϊκή καριέρα, ιδιαίτερα δηλαδή στην εκπαίδευση, κάτι το οποίο μας θίγει και ως ευρωπαϊκή αντίληψη και κυρίως ως φίλο. Η δεύτερη ενότητα αφορά στα μέτρα, στα θετικά μέτρα τα οποία μπορούμε, με τα οποία μπορούμε σε αυτό το πρόβλημα να βάλουμε ε, σημαντικά ε, βήματα, να κάνουμε σημαντικά βήματα. Το λέω αυτό γιατί γνωρίζετε όλοι ότι αυτές οι εκθέσεις πολλά χρόνια απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το γεγονό ότι την απασχολούν ακόμη μα προσβάλλει ω γυναίκε και ω ευρωπαίου πολίτε Και μα προσβάλλει γιατί είναι αδιανόητο στην εποχή που ζούμε να υπάρχουν ακόμη διακρίσει. και μάλιστα σε επίπεδο ανισότητος εκεί όπου η γυναίκα έχει αποδείξει χωρίς να χρειάζεται να το αποδεικνύει πάντα, αλλά το έχει αποδείξει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στο έπακρο σε όποιο ρόλο αναλαμβάνει. Τα θετικά μέτρα αφορούν στις νομοθεσίες των κρατών μελών. Υπάρχουν νομοθεσίες οι οποίες πραγματικά δεν βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν σε άλλες χώρες που είναι πιο προηγμένες. Καλό θα είναι λοιπόν εφ' εξής, να ακολουθηθεί μια, μια ευρωπαϊκή στρατηγική που με έναν τρόπο να εναρμονίζει τις νομοθεσίες σε θετική κατεύθυνση. Παράλληλα όμως με την νομοθεσία, δηλαδή τις νομοθεσίες στα επιμέρους κράτη-μέλη, αλλά και ένα νομοθετικό μια νομοθετική ομπρέλα που θα μπορεί να εκπονήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή που είναι νομοθετικό σώμα, ε, υπάρχουν και οι εκστρατείε ενημέρωσης. Δηλαδή ουσιαστικά αν δεν υπάρχει η ενημέρωση είτε των εμποδίων που υπάρχουν στην εξέλιξη των γυναικών, στην εκπαίδευση και στην έρευνα, είτε των τρόπων με τον οποίο μπορούν να έρθουν αυτά τα εμπόδια, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Στην τρίτη ε, κατηγορία, η οποία συνδέεται και με αυτή τη δεύτερη, αναφέρομαι στις παροχές και τα κίνητρα από τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα ε, στις γυναίκες της παραγωγικής ηλικίας μετά τη μητρότητα. Εκεί πραγματικά, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, και παίρνω ένα παράδειγμα από τη χώρα μου, έχει σημασία αυτό, βλέπουμε πολλές γυναίκες και μάλιστα υψηλών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων να χάνουν την εργασία τους όταν εκ του νόμου που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατοχυρώσει νομοθετικά το δικαίωμα της απουσίας συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα από την εργασία, αυτό ουσιαστικά να στρέφεται εναντίον τους, να στοχοποιούνται και να θεωρείται ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν διότι δεν έχουν ενημερωθεί, ε, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του τομέα στον οποίο έχουν αναλάβει. Αυτό βέβαια είναι πρόσχημα, διότι ε, δυστυχώς και εδώ ρατσιστικά ε, λειτουργούν ορισμένοι τομείς, υποτιμούν την ε, ανάγκη να ε, πλαισιώνονται αυτοί οι τομείς από γυναίκες. Ε, στην τέταρτη κατηγορία προτείνουμε κάποιες αλλαγές στους τομείς ορίζων 2020 και στον ευρωπαϊκό τομέα έρευνας της Επιτροπής και μάλιστα οι αλλαγές είναι, περιγράφονται. Τώρα σας κάνω μια έτσι συνολική αναφορά. Μετά θα ακούσω και τις παρατηρήσεις σας και εννοείται ότι έχουμε σε εξέλιξη και σε επίπεδο τροπολογιών αλλά εδώ θα ήταν χρήσιμο κάτι το οποίο ε, πρέπει να παρακολουθείτε κατέτος, δηλαδή στατιστικές. Οι στατιστικές να μας λένε σε ποια κράτη-μέλη παρουσιάζουμε οι θέσεις και εξάρσεις του φαινομένου και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα και ιδιαίτερα στα ε, πανεπιστήμια ας πούμε και στα κέντρα έρευνας όπου πραγματικά υπάρχει ουσιαστική ε, υποεκπροσώπηση των γυναικών, ενώ αντίθετα δεν συμβαίνει αυτό τουλάχιστον στη χώρα μου στο δικοστικό κλάδο. Σας λέω ας πούμε μια άλλη ε, παράμετρο και ίσως εκεί διότι οι γυναίκες που επιλέγουν το δικοστικό κλάδο ε, εστιάζουν πάνω στην σιγουριά ενός μισθολογικού καθεστώτος το οποίο αναβαθμίζεται στη δικαστική εξουσία αλλά αυτό δεν θα πρέπει να είναι το κίνητρο. Το κίνητρο είναι πάντοτε και η δημιουργία στη γυναίκα και το έχει αποδείξει. Ε, ακολούθως, ε, στο, στην επόμενη κατηγορία, πέμπτη, ε, θα πρέπει να αναλύσουμε τα θετικά βήματα προόδου. Δηλαδή μια εκτεταμένη στρατηγική η οποία ε, θα, θα αναφέρεται στο κατά πόσο μεθοδευμένα και χωρίς ε, αποκλήσει θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά να βοηθήσει τα κράτη-μέλη έτσι ώστε η εναρμόνιση της νομοθεσίας την οποία αναφέρθηκα πριν θα έχει να κάνει και με μια μεθοδευμένη αλλαγή νοοτροπίας. Μην ξεχνάμε ότι τα δύο φυτόρια όπως συνηθίζω να λέω και όταν έκανα πρακτική δικηγορία το έλεγα που είναι η οικογένεια σε πρώτο επίπεδο και η παιδεία σε δεύτερο, ιδιαίτερα εκεί όπου διαμορφώνεται ο χαρακτήρας των προσωπικότητων, στην εφηβεία, στη μέση εκπαίδευση, αν έχει οργανωμένα προγράμματα, οργανωμένα μαθήματα και ειδικού εκπαιδευτέ, οι οποίοι θα καθοδηγούν τα παιδιά να αντιλαμβάνονται ότι η ισότητα δεν είναι μία αφηρημένη έννοια ή μία διεκδίκηση των γυναικών, είναι μία αξία που αφορά στους πολίτες που γεννήθηκαν άνθρωποι και απλώς διακρίνονται σε δύο φύλλα από τη φύση. Αλλά ως προς τα δικαιώματά τους δεν θα έπρεπε ποτέ να συζητάμε για διακρίσεις. Αυτό είχα την τιμή να το πω και στην Ολομέλεια όταν το η άλλη έκθεση, παράλληλη έκθεση, διότι δυστυχώς οι διακρίσεις δείχνουν παγιωμένες στερεότυπα και νοοτροπίες οι οποίες παρά τις προσπάθειες όλων μας δεν έχουν αλλάξει και δεν έχουν αλλάξει σε τέτοιο σημείο που να μην συζητάμε τέτοια θέματα. Ελπίζω μετά από χρόνια να φτάσουμε σε αυτή την εξέλιξη. Το ελπίζω τουλάχιστον. Ε, πέραν των, προγραμμάτων που, στα οποία αναφέρομαι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στη μέση, στην ε, μέση εκπαίδευση αλλά και στην οικογένεια σε επίπεδο καθοδήγησης, εκτιμώ ότι σε κάθε κράτος μέλος με τη δική μας την προτροπή ως Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να εκπονηθούν εκστρατείες ενημέρωσης σε επίπεδο ημερίδων, διημερίδων, ειδικών φόρουμ, φόρα δηλαδή λέγονται αυτά στο πληθυντικό, όπου πραγματικά θα υπάρχει αυτό το αντικείμενο, όχι όμως σαν ένα αντικείμενο ε, φιλολογικού διαλόγου ή εκπαιδευτικού διαλόγου, θα υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένες κατευθύνσεις, εφικτά μέτρα, τα οποία μπορούν και θα πρέπει να με έναν τρόπο πιεστικό να επιβάλλονται. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Δηλαδή παράλληλα η νομοθετική εξουσία με την εκπαίδευση σε σύνολο, σε θετική κατεύθυνση, θα μπορεί να παραγάγει ε, πολύ ουσιαστικά αποτελέσματα. Και τελειώνοντας, ε, κλείνοντας, το τελευταίο κεφάλαιο της έκθεσης τονίζουμε την ανάγκη της συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων ε, ε, φορέων. Το λέω διότι παρατηρούμε ότι ειδικά ας πούμε ε, στην έρευνα, στα διοικητικά συμβούλια, στα επιστημονικά ιδρύματα, όχι μόνο υποεκπροσωπούνται οι γυναικείες παρουσίες, αλλά σε πολλά από αυτά δεν υπάρχουν καθόλου. Αυτό ε, ε, θα μου επιτρέψετε να πω ότι πέραν της νοοτροπίας είναι ανησυχητικό. Και το λέω ανησυχητικό, παίρνω παράδειγμα πρόσφατα, ξέρετε ότι βραβεύθηκε με ε, τον Νόμπελ Ιατρικής ο βιολόγος Tim Hunt, ο Εγγλέζος βιολόγος Tim Hunt. Ένας άνθρωπος 72 χρονών που θεωρήθηκε ότι εκφράζει ανοιχτούς ορίζοντες πέραν της επιστήμης του, αυτός ο άνθρωπος δήλωσε δημόσια ότι είναι σοβινιστής, και ότι ειδικά στα κέντρα έρευνας δεν πρέπει να υπάρχουν γυναίκες, διότι είτε τις ερωτεύεσαι και χρησιμοποιείς προσωπικές σχέσεις, είτε όταν ε, τολμήσεις να τους υποδείξεις ένα σωστό δρόμο και να κάνεις παρατήρηση, βάζουν τα κλάματα. Αυτό αντιλαμβάνεστε από έναν νομπελίστα, ο οποίος βέβαια μετά επικρίθηκε και από όλα τα επιστημονικά φόρα και από μεμονωμένες προσωπικότητες, αλλά δεν είναι ένα, μία εξαίρεση που θα λέγαμε ότι είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Διότι δεν είναι τυχαίο ότι είναι νομπελίστας, δεν είναι τυχαίο ότι είναι ένας πνευματικός άνθρωπος. Αν λοιπόν, σαν και αυτόν, υπάρχουν κάποιοι άλλοι που απλώς δεν εκφράζονται δημόσια για να επικριθούν, αλλά ουσιαστικά ε, απαρτίζουν μια κατηγορία εσφαλμένης και νοσηρής αντίληψης, σημαίνει ότι είναι ριζωμένες αυτές στην κοινωνία μας οι νοοτροπίες και η εκρίζωσή τους μπορεί μόνο με μεθοδευμένες συστηματικές συνειδητές προσπάθειες να μπορέσει να παραγάγει αποτελέσματα. Αυτό το έφερα όχι για να στιγματίσω το συγκεκριμένο άνθρωπο, διότι έχει στιγματιστεί από τις δηλώσεις του και από όλες αυτές τις ε, αποδοκιμασίες που εισέπραξε. Αλλά δείχνει μια παθολογία και είμαι υποχρεωμένη να τη συμπεριλάβω ε, για την ολοκλήρωση του σκεπτικού μου. Ε, τελειώνοντας να πω λοιπόν ότι αυτοί είναι οι, οι βασικοί άξονες της εκθέσεως. Εννοείται ότι μέχρι την ημερομηνία που έχει δοθεί οι τροπολογίες, οι παρατηρήσεις και οι εισηγήσει όλων σας θα ληφθούν υπόψη ε, και θα είναι και πολύ επιβοηθητικές για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε μια έκθεση που δεν θα είναι μια έκθεση θεωρητικού περιεχομένου αλλά θα προτείνει συγκεκριμένες δράσεις και αφού σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας, να πω ότι θα είμαι στη διάθεσή σας πέραν των emails που μπορείτε να μας στείλετε ε, και προσωπικά εγώ, σε οποιαδήποτε συναντήσεις θα θελήσετε να έχουμε και προσωπικά και με τους συνεργάτες μου και σε τεχνικό επίπεδο. Και να ευχαριστήσω και πάλι. Thank you, Mr. Σας ευχαριστούμε κυρία Βόζεμπεργκ. Μας κάνατε μια παρουσίαση πολύ άρτια και εμπεριστατωμένη ενός θέματος που θα απασχολήσει την Επιτροπή και μας ενισχύει και όλα. Γύρω συζητήσαν τώρα. Πρώτα θα δώσω το λόγο στους και ηγητές από τις διάφορες ομάδες. Πρώτα η κυρία Νταντζίλα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τη συνάδελφό μας, Ελίζα ε, Βόζεμπερκ, για την έκθεση την οποία σήμερα συζητούμε. Όπως ε, πολύ εύστοχα είπε η κυρία η συγγήτρια εκπροσωπούνται οι γυναίκες σε πολύ σημαντικούς τομείς της κοινωνίας, της επιστήμης, της έρευνας ε, και στη λήψη των αποφάσεων και γενικότερα σε πολλά υψηλά επίπεδα που λαμβάνονται αποφάσεις. Γενικά, θα πρέπει να πούμε ότι οι γυναίκες είναι όλο περισσότερο παρούσες στη διοίκηση και στην παροχή υπηρεσιών. Αλλά ταυτόχρονα διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Είναι περιορισμένη η παρουσία τους στις υπηρεσίες σε θέσεις χαμηλών προσόντων και σε χαμηλή ε, ιεραρχική βαθμίδα. Οπότε οι γυναίκες δεν είναι παρούσες στην ε, ε, ζωή, στο εργασιακό βίο ε, εξίσου με τους άνδρες. Ε, με πολύ πιο επισφαλή θέση, πολύ ωραία το εξήγησε η κυρία Βόζεμπερ για γυναίκες που γεννούν και στη συνέχεια χάνουν τη δουλειά τους ακριβώς επειδή γέννησαν. Και οι διαφορές οι είναι πολύ μεγάλες και το χάσμα και η ψαλίδα διευρύνεται περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα παρά στο δημόσιο. Ε, έχουμε στατιστικές τις οποίες παρουσιάζει και η ίδια η συγγήτρια που δείχνουν ότι χιλιάδες νέες γυναίκες ε, που ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την επιστήμη τους ε, συναντούν αόρατους φραγμούς και εμπόδια. Στη στρατηγική για το 2020 έχουμε στόχο να προωθήσουμε την παρουσία των γυναικών στην επιστήμη χωρίς αποκλεισμούς. Σήμερα περισσότερο από ποτέ ο κόσμος έχει ανάγκη την επιστήμη αυτή. Και όπως πολύ ωραία λέγει η έκθεση, και οι επιστήμες χρειάζονται περισσότερο τις γυναίκες που ενέχονται με πολύ πάθος, με ζέση, με ενθουσιασμό. Οι ερευνήτριες είναι γυναίκες ε, έξυπνες ε, που αποφασίζουν να αφοσιωθούν, να αφιερώσουν τη ζωή τους στην έρευνα. Στις σύγχρονες ερευνητικές ε, προκλήσεις. Ως και συγγήτρια των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα καταθέσω και τροπολογίες ε, προς την κατεύθυνση αυτή για να επιμείνουμε ακριβώς όπως είπε και η κυρία Βόζεμπεργκ είναι πάρα πολύ ωραία, θα πρέπει να επικεντρωθούμε ακριβώς σε αυτό. Συγκεκριμένες προτάσεις να κάνουμε και όχι γενικά σχόλια και θεωρητικές εκτιμήσεις για να συμμετέχουν περισσότερο γυναίκες σε όλα αυτά τα θέματα. Θα ακούσουμε μεγάλη προσοχή ε, όλους τους συναδέλφους και είμαι βέβαια ότι μαζί με την εισηγήτρια θα βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για να αντανακλά την ε, πραγματικότητα, η έκθεση και να βοηθάει και τις γυναίκες. Ευχαριστώ Εγώ τους φιλελευθέρους. Thank you very much, uh, Madam Chair. I would also like... Κύριε Μίλα, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω και να συγχαρώ καταρχάς την εισηγήτριά μας, κυρία Βόζεμπερκ, ε, για το μέχρι τώρα έργο της. Νομίζω ότι το σχέδιο έκθεσης όπως περιέγραψε η κυρία Βόζεμπερκ, αντιμετωπίζει όλες τις μεγάλες προκλήσεις των γυναικών ακριβώς όταν θέλουμε να ακολουθήσουμε επιστημονική σταδιοδρομία. Και, ε, αυτό υπάρχει σε πολλούς τομείς. Ε, και υπάρχει το θέμα ε, της συμφιλίωσης του επαγγελματικού με τον ιδιωτικό βίο και κάποια άλλα θέματα πιο ειδικά. Θα ήθελα εγώ να ενισχυθούν τα κεφάλαια που διαπραγματεύονται πιο συγκεκριμένα προβλήματα. Τι εννοώ, εννοώ τους φραγμούς στην ε, χρηματοδότηση για την έρευνα και όπως είπε προηγουμένως και συνάδελφος των σοσιαλιστών, το χάσμα, το μισθολογικό. Αυτά τα οικονομικά ε, ζητήματα μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά ε, τις επιλογές των γυναικών, αν θα επιλέξουν μια τέτοια καριέρα δηλαδή όχι. Και χρειάζονται μεγάλα βήματα στον επιστημονικό τομέα προς την ισότητα, και δεν είναι μόνο απαραίτητο αυτό, είναι και δυνατό. Το είπε και η κυρία Βόζεμπερτ ότι υπάρχουν άνθρωποι μέχρι και νομπελίστες που εκφράζουν τέτοιες απόψεις. Τελικά είναι και σεξιστές μέχρι και ρατσιστές. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να μας αποτρέπει, να μας εμποδίζει από το να κάνουμε τη δουλειά μας και να στρέφουμε τα πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Από τους Πρασίνους, ο κύριος Σεμπαστιάν. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Βόζεμπερκ. Νομίζω πως η έκθεση είναι πολύ καλά, είναι πολύ καλή και πως όλες οι διεκδικήσεις ε, που έχουμε, έχουμε κάνει σε αυτήν τον τομέα ε, αναφέρονται στην έκθεση αυτή. Τώρα, αλλά η κατάσταση είναι πολύ πιο σκληρή ε, για τις γυναίκες. Δεν ξέρω σε άλλες χώρες, αλλά στην Ισπανία γενικά η φοιτήτριε γυναίκες ε, έχουν καλύτερες ε, ειδικότητε, λαμβάνουν καλύτερε ε, και στον τομέα των εργασιακό αλλά και στον ερευνητικό και επαγγελματικό. Εμείς θα, δουλέψουμε πάνω σε κάποιες τροπολογίες με τρεις, τρεις βασικούς άξονες. Το πρώτος είναι το θέμα της συμβατότητας της επαγγελματικής και της οικογενειακής εργασίας. θα πρέπει ζωή, συγγνώμη, θα πρέπει να στηρίξουμε τα μέτρα προκειμένου οι γυναίκες να μπορέσουν να συνδυάσουν την οικογενειακή ζωή με την επαγγελματικό βίο. Θα πρέπει να καταβάλουμε επίση προσπάθεια προκειμένου να απαιτήσουμε από τους άντρε οι οποίοι και αυτοί θα πρέπει να ενταχθούν και να συμμετάσχουν στην οικογενειακή ζωή έτσι ώστε οι γυναίκε να έχουν μεγαλύτερο χρόνο ελεύθερο και να αναλάβουν και οι άντρε τι ε, ευθύνε του. Να ενταχθούν λοιπόν σε αυτόν τον οικογενειακό βίο που σε πολλέ περιπτώσει ε, αυτό δεν συμβαίνει. Ε, και έτσι πολλές εργασίες οικογενειακές αναλαμβάνονται, αναλαμβάνονται από τις γυναίκες. Θα πρέπει λοιπόν να ενταχθούν και οι άντρες σε αυτές τις εργασίες. Οι γυναίκες λοιπόν θα πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα με τους άνδρες να ενταχθούν δηλαδή οι άνδρες στην οικογενειακή ζωή και τη φροντίδα της οικογένειας, η οποία θα πρέπει να είναι αποκλειστική μέρη της γυναίκας. Θα πρέπει να διευκολύνουμε την συμβατότητα με την ε, οικογενειακή ζωή και την επαγγελματική. Επαναλαμβάνω ότι αυτό ε, θα αποβαίνει συχνά εις βάρος της γυναίκας ε, και το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να δείξω είναι κάτι που έτυξε ήδη η συγκήτρια, το θέμα των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Δηλαδή, ο διαχωρισμός μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα είναι θεωρητικής περισσότερο διότι το μεγαλύτερο κομμάτι της έρευνας ε, λαμβάνει και δημόσια στήριξη, κρατική επιχορήγηση. Θα πρέπει λοιπόν οι γυναίκες να μπορούν να εποφελούνται από αυτήν την ε, κατάσταση. Να μπορούν οι γυναίκες λοιπόν να εποφελούνται από αυτές τις ε, εξελίξεις. Φυσικά στον ιδιωτικό κλάδο είναι πιο δύσκολο να ενταχθούν οι γυναίκες ε, στον τομέα της έρευνας. Και ένα τρίτο σημείο που θα ήθελα να αναφερθώ είναι το επαγγελματικό αποτέλεσμα. Αυτό το βραβείο Νόμπελ που το οποίο ανέφερε η συγγήτρια είπε ότι είναι φυσιολογικό άτομα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό το πρόσωπο. Έχει σίγουρα διάφορα προβλήματα. Το... Σε πολλές περιπτώσεις λοιπόν τα περιεχόμενα της έρευνας είναι, έχουν καθαρά ανδρικό χαρακτήρα. Η μη ένταξη των γυναικών στον τομέα της έρευνας έχει ως αποτέλεσμα όπως σε ζητήματα όπως τα ιατρικά και που αφορούν κλάδους στους οποίους εμπλέκονται οι γυναίκες ε, δυστυχώς όμως υπάρχει μεγαλύτερη ανδρική παρουσία οι γυναίκες παραμένουν εκτός σε πολλές περιπτώσεις πάνω σε αυτά θα πρέπει να δουλέψουμε και τονίζω ότι το σημείο κίνησης είναι πάρα πολύ καλά και συγχαίρω την εισηγητή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σεμπαστιά. Πριν δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζήτησε το λόγο κυρία Μπέτιο. Παρόλο που αργότερα θα μας παρουσιάσει μια μελέτη, ζήτησε το λόγο και τώρα. Μια ναι, και έχουμε λίγο χρόνο, θα της δώσω το λόγο πείτε μας δύο λόγια για και μετά μπορείτε να εκφέρετε και τη γνώμη σας. Um, uh, Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δώσατε την ευκαιρία για να κάνω μια άτυπη ε, παρέμβαση γιατί για άλλο λόγο βρίσκομαι εδώ, θα σας παρουσιάσω αργότερα τη μελέτη. Θα ήθελα απλώς ε, να επιστήσω την προσοχή των μελών της Επιτροπής Γυναικών σε κάτι που συμβαίνει σε σχέση με τον ορίζοντα 2020. Από ό,τι φαίνεται, με βάση ε, διακεκριμένους επιστήμονες που εξετάζουν τα θέματα της χρηματοδότησης, φαίνεται ότι στη χρηματοδότηση το κριτήριο του φύλου δεν λειτουργεί αρκετά καλά σε ό,τι αφορά την επιλογή σχεδίων και προγραμμάτων που πραγματικά ε, λαμβάνουν υπόψη και το θέμα των φύλων. Και δεν μιλώ μόνο για τη σταδιοδρομία, αλλά τη συνεκτίμηση του φύλου σε θέματα επιστημονικά, που είναι εξίσου αν όχι περισσότερο σημαντικό θέμα. Σε αυτό το ζήτημα θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας και σε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στο τεύχος 15 του Science and Technology. Μπορείτε να το έχετε διαβάσει. Εκεί γίνεται ανάλυση της παρούσας κατάστασης ε, και το τι με λιγενέστε. Γίνεται μια επίσημη προσπάθεια, μια επίσημη απόπειρα, στην οποία συμμετέχω και εγώ, από μια ομάδα που προσπαθεί να ασκήσει πίεση και να ληφθούν υπόψη τα να ληφθεί υπόψη το θύλο και να αλλάξουν τα κριτήρια στον επόμενο γύρο. Και σας ευχαριστώ για το λεπτό που μου δώσατε. Ευχαριστούμε κυρία Βερτιόλα για την ε, πληροφορία που μας δώσετε, να είστε βέβαιοι ότι θα τη λάβουμε υπόψη και στο δικό μας έργο, στις δικές μας εργασίες. Θα δώσω τώρα το λόγο στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Γουίλης Μάτσης. Σας ακούμε. Σας ευχαριστώ. Ονομάζομαι Βίλης Ματσίκη και είμαι ματάρχης στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογικής, ανάπτυξη και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, μάλλον, για θέματα φύλου. Θα ήθελα να χαιρετήσω την έκθεση αυτή για τις γυναίκες στην επιστήμη και στον πανεπιστημιακό κλάδο, γιατί πραγματικά με μεγάλη οξυδέρκεια μιλώ όχι μόνο για τις ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων, αλλά επισημαίνει τις ιδιαιτερότητες ε, της έρευνας και της καινοτομίας ε, σε θέματα δημοσιεύσεων, ε, λήψη αποφάσεων, πρόσβαση στη χρηματοδότηση και ούτω καθεξής. Η στρατηγική που αναπτύσσουμε τώρα από κοινού με τα κράτη-μέλη περνάει από τις άμεσες ενισχύσεις στις γυναίκες επιστήμονες, που είναι σημαντική, αλλά πρέπει να κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς θεσμικές αλλαγές στην οργάνωση, στη διοργάνωση της έρευνας, ώστε να προσαρμόσουμε κάποιες πρακτικές αλλά και κάποιες νοοτροπίες στις νέες συνθήκες, να ξεπεράσουμε κάποια στερεότυπα στην οργάνωση της έρευνας. Και αυτή γίνεται μια απόπειρα και στα κράτη-μέλη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Χώρου. Και τελευταία πρωτοβουλία ήταν η απόφαση του Συμβουλίου του περασμένου Μαΐου για τη θέσπιση ενός οδικού χάρτη στα κράτη-μέλη, προκειμένου να καταρτιστούν εθνικά σχέδια δράσης και στρατηγικές σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι, το, μέχρι τα μέσα του 2016. Οπότε πραγματικά η έκθεση είναι πολύ επίκαιρη. Υποβάλλεται την κατάλληλη στιγμή και θα στηρίξει τις αντίστοιχες προσπάθειες των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ και για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση θα ξαναδώσουμε το λόγο στην εισηγητριά μα την κυρία Βόζεμπερκ. Κυρία Πρόεδρε, να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις ε, συνεισηγητές γιατί θεωρώ ότι η εισήγηση είναι διαδραστική πάντοτε όταν συνδράμουν το έργο μιας έκθεσης. Όλοι έχουμε τον ίδιο βαθμό ευθύνη και την ίδια αξία συμμετοχής με χαρά μου άκουσα και όλες τις ε, συναδέλφους και τον μοναδικό άνδρα εισηγητή των Πρασίνων, ο οποίος είπε και πολύ σημαντικά πράγματα, διότι αναφέρθηκε, κάνω ειδική αναφορά, διότι προς τιμήν του αναφέρθηκε στην ανισότητα που υπάρχει ακόμη και στην οικογένεια σε σχέση με τους ρόλους που έχουν παραδοσιακά απονεμηθεί στον άντρα και στη γυναίκα με αποτέλεσμα αυτό να ενισχύει και να εμπλουτίζει πολλές φορές εσφαλμένες νοοτροπίες χωρίς να σημαίνει ότι ποτέ διεκδικήσαμε εμείς οι γυναίκες να πάρουμε ρόλο που ανήκει σε, άλλο, σε άντρα αλλά αυτά τα καθορίζει η φύση δεν τα καθορίζουν οι νοοτροπίες οι νοοτροπίες αλλάζουν Επίσης ε, να ευχαριστήσω και τη συνάδελφο των φιλελευθέρων ε, η οποία επεσήμανε την ανάγκη για την ε, εξίσωση στη μισθολογική τη μισθολογική εξίσωση σε γυναίκες οι οποίες κατέχουν τα ανώτατα αξιώματα και δεν αμείβονται με τον ίδιο τρόπο, διότι αυτό παρά το γεγονός ότι και στα κράτη-μέλη έχει γίνει μεγάλη εξέλιξη από ό,τι έχω διαβάσει και μελετήσει στις μισθολογικές αναφορές, δεν εφαρμόζεται ο νόμος με αποτέλεσμα να υπάρχουν ε, σωρία αγωγών οι οποίες προσφεύγουν στα δικαστήρια προκειμένου να ε, ε, διεκδικήσουν το αυτονόητο. Επίσης να ε, πήγα λίγο αντίστροφα τη συνάδελφο από τους σοσιαλιστές που μίλησε για την ανάγκη της εξειδίκευσης των δράσεων. Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη. Ακριβώς αυτό είναι ο ρόλος μας, γιατί διαφορετικά η έκθεσή μας δεν θα έχει ούτε δυναμική ούτε και πιεστικό μοχλό, μπορούμε να πούμε, αν δεν εξειδικεύει τις δράσεις. Ε, πολύ σωστή ήταν και η παρατήρηση ε, εννοείται της ε, κυρίας Σουήλης με ευχαρίστησε το γεγονός ότι επεσήμανε την επικαιρότητα της έκθεσης αυτής που θα μπορούσε να βοηθήσει εφόσον το Συμβούλιο μαζί με την Επιτροπή εκπονεί δράσεις που να ε, βοηθούν στην κατεύθυνση και των οικονομικών ισοτήτων αλλά κυρίως της προτροπής προς τις γυναίκες να μπορούν να δικαιούνται, να αξιώνουν αυτό το οποίο δικαιούνται, δηλαδή να ασκούν ουσιαστικά τα δικαιώματά τους στην ανώτατη εκπαίδευση και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Και ε, θα έπρεπε να είναι δίδαγμα, και τελειώνω με αυτή την παρατήρηση κυρία Πρόεδρε, θα έπρεπε να, να μας γίνεται παράδειγμα το γεγονός ότι στα ελεύθερα επαγγέλματα οι γυναίκες, μπορώ να σας πω ότι σε πολλά κράτη-μέλη πρωταγωνιστούν. Και εκεί διότι δεν υπάρχουν ούτε μοχλή αξιολόγηση που μπορεί να μην είναι αντικειμενική, ούτε κάποιοι προωθητικοί μηχανισμοί που να εισάγουν ανισότητες. Είναι το ελεύθερο πεδίο όπου οι άνθρωποι άντρες γυναίκες μπορούν να αποδείξουν τις ικανότητές τους και να αντέξουν να έχουν και πολλές, πολλούς ρόλους όπως οι γυναίκες που από τη φύση τους εκ των πραγμάτων επομίζονται και κάποια ειδικά καθήκοντα τα οποία βεβαίως και ποτέ δεν θέλησαν να απεμπολίσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Βόζεμπεργκ. Η εργασία λοιπόν θα συνεχιστεί σε συνεργασία με τους γιώδεις συζητητές και με βέβαιη πως το αποτέλεσμα θα είναι διότι το θέμα έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για τις γυναίκες αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση το σύνολό της και για όλους τους πολίτες. Περνάμε στο επόμενο σημείο, υπερασμό 15 σχετικά με την αποστολή στη Νέα Υόρκη. Έχετε στα έγγραφά σας μια έκθεση από που μπορείτε να γνωρίσετε τόσο τη στη διάταξη όπως και τα αποτελέσματα αυτών των συνεδριάσεων που είχαμε ως εκ τούτου απλά προς ενημέρωση και να περάσουμε στο επόμενο σημείο της μεριστίας διάταξης που αφορά στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ανθρωπιστικής ε, βοήθειας ε, υπάρχει μια νομοδότηση της οποίας η συγγήτρια είναι η κυρία Χέιντ. Θα της δώσω το λόγο λοιπόν για να μας ε, κάνει μια εισαγωγή στην συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. σε naturkatastrofer. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, στο θέμα των συγκρούσεων των θεμηνιών ε, κυριαρχεί αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ε, ε, κυβερνήσεις από τον κόσμο ολόκληρο αλλά και ΜΚΟ και θύματα ε, θεομηνιών θα συνεδριάσουν του χρόνου το Μάιο στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ ιδιαίτερη σημασία έχει και το ζήτημα της σεξουαλικής βίας ή της σεξουαλικής εκμετάλλευσης σε σχέση με θεομηνίες και καταστροφές. Διότι πάρα πολύ συχνά ε, οι ε, πιο ευάλωτοι πλήττονται από όλες τις καταστροφές και τις σειράξεις και ακόμα περισσότερο από αυτό. Σε πολλές περιφέρειες του κόσμου και χώρες, κυρίως γυναίκες και παιδιά ε, που είναι θύματα καταστροφών και θεομηνιών, πέφτουν και θύματα καταπίεσης και ανισοτήτων. Τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε την ευκαιρία να ε, εντείνουμε την πίεση που ασκούμε στις κυβερνήσεις παγκοσμίω, αλλά και στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που ε, δραστηριοποιούνται στην πολιτική προστασία και στην αντιμετώπιση των θεομηνιών για να συμπεριλάβουν και το gender mainstreaming. Γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ για την ευκαιρία που έχουμε να συζητούμε αυτό το θέμα και που ορίστηκα εγώ εισηγήτρια για τη συγκεκριμένη έκθεση. Ελπίζω από κοινού να καταλήξουμε σε μια γνωμοδότηση λογική. Πρόκειται, είτε πρόκειται για τη διατήρηση της ειρήνης είτε για ε, τμήματα που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές όλοι οι εργαζόμενοι και οι διασώσεις θα πρέπει να γνωρίζουν τις ε, κατάλληλες συνθήκες, τις κατάλληλες εργασίες για να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες που προκύπτουν κάθε φορά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να μπορούμε να βοηθήσουμε με αποτελεσματικό τρόπο τους πλέον εκτεθειμένους, διότι βία η οποία βασίζεται στο φύλλο και αφορά οικονομική, φυσική και αλλά και σεξουαλική βία δεν είναι ένα νέο φαινόμενο και δεν περιορίζεται φυσικά σε ορισμένες περιοχές του κόσμου. Όλοι βλέπουμε από τις πληροφορίες που φτάνουν από τον κόσμο είναι ότι υπάρχουν πολλές φορές ε, ότι όπου οι γυναίκες ε, πλήττονται από την Αφρική, Λατινική Αμερική. Συχνά λοιπόν βλέπουμε ε, τρομερά δείγματα βίας και αυτό αφορά σίγουρα την ε, διαφορά ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Υπάρχει λοιπόν μια συστηματική θα έλεγα βία κατά των γυναικών και αυτό οδηγεί σε ε, τις γυναίκες να βρίσκονται σε πιο υποβαθμισμένες συνθήκες ε, σε ό,τι φορά τώρα τη σεξουαλική βία και ιδιαίτερα τους βιασμούς διαπιστώνουμε ότι ο βιασμός χρησιμοποιείται ως συστηματικό μέσο ε, κατά των γυναικών αλλά και των παιδιών πολλές φορές. Είναι απαραίτητο να παρέμβουμε κατά αυτής της πραγματικότητας και τώρα έχουμε δυνατότητα να ασκήσουμε πίεση στα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή τα άτομα τα οποία ασχολούνται σε αυτούς τους τομείς προκειμένου να λάβουν υπόψη την ισότητα των φύλων. Χρειάζεται να μην ξεχνάμε πως ε, αυτή είναι μια προοπτική ε, της ε, μορφής bottom-down, δηλαδή από την κορυφή προς τη βάση. Θα πρέπει να γνωρίζουμε επίσης ότι αυτό αφορά και όλους όσοι βίασαν ε, παιδιά. Ας δούμε τι συνέβη στην ε, Κεντρική Αφρική, στη Δημοκρατία της Κεντρικής Αυτά τα πρόσωπα τα οποία στέλνει ο ΟΗΕ είναι κατάλληλα καταρτισμένα, αλλά θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα καταρτισμένα στην ε, γυναικεία στην στάση που θα πρέπει να, να οποία πρέπει να, με την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τις γυναίκες οι οποίες ε, έχουν δωρήσει πολλές μορφές βίας στις περιοχές αυτές. Πρέπει λοιπόν να ασκήσουμε περισσότερη πίεση και σε κυβερνητικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο οργανώσεων που, εργάζονται επιτοπίως θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι όσοι αντιμετωπίζουν έκτακτες καταστάσεις να προστατεύονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Αυτά και περιμένω τις, ε, το σχολιασμό σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στις παρεμβάσεις ε, των ε, εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων. Κύριε Ζαμπόρσκα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Χέντ την εισηγήτριά μας, για την παρουσίαση του εγγράφου που μας έκανε. Ε, μας κάλυψε σε όλα τα σημεία κυρία Χέντ Ήταν πραγματικά πολύ διεξοδική η ενημέρωση που μας έκανε και πιστεύω ότι η Επιτροπή των Γυναικών θα συμβάλλει στην διαμόρφωση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν ώψη της διάσκεψης της Κωνσταντινούπολης. Θα ήθελα να σταθώ σε κάτι που ήδη αναφέρατε και που είναι πραγματικά αποτρόπαιο και φρικιαστικό. Είναι σκανδαλώδες ότι επίσημο προσωπικό, μία επίσημη μονάδα ανθρωπιστικής βοήθειας ε, διεθνούς οργάνωσης κάνει κατάχρηση της θέσης της ε, και ανταλλάσσει καλλιτικά ή τροφή για σεξ. Είναι πραγματικά έσχος. Και σε κάποιες χώρες της Μέσης Ανατολής ε, ή της Αφρικής μερικές φορές στρατιώτες χρησιμοποιούν το βιασμό ως όπλο και το στυλιτεύουμε βέβαια και το καταδικάζουμε, αλλά εδώ πρόκειται για εμπόλεμη σύραξη. Δεν το δικαιολογώ, αλλά εδώ βλέπουμε επίσημα στρατεύματα ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανώσεων που αποδίδονται σε τις πρακτικές. Αυτό και αν είναι απαράδεκτο και επονίδιστο. Οι γυναίκες είτε σε εμπόλεμες σειράξεις σε αναπτυσσόμενες χώρες, είτε σε οποιοδήποτε θεομηνία ή φυσική καταστροφή, οι γυναίκες είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο και υποφέρουν. Είναι υπεύθυνε και για τις οικογένειές τους και φέρνουν όλο το βάρος και να κάνει κανείς κατάχρηση αυτής της κατάστασης και της αδυναμίας του είναι πραγματικά ε, ντροπή και παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Σας ευχαριστώ κύριος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτριά μας. Σε γενικές γραμμές ε, συμφωνώ και θέλω να σας ευχαριστήσω ε, για το γεγονός ότι επιλαμβάνεστε του θέματος Αυτό Είναι πολύ σημαντικό. Είναι σκάνδαλο αυτό που ακούμε καθημερινά ε, ότι γίνονται επιθέσεις, πώς να το πω τώρα, άνθρωποι που πρέπει κανονικά να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους σε περιοχές που έχουν ε, πληγή από πολέμους ή καταστροφές και τι κάνουν σε ανυπεράσπιστες γυναίκες και παιδιά. Αλλά είναι γενικότερα πολιτισμικό το πρόβλημα. Έχουμε φτάσει μέχρι το φεγάρι και μέχρι τους βυθούς του ωκεανού. Στέλνουμε ε, ε, δορυφόρους στα όρια του διαστήματος και του σύμπαντος, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουμε μεταξελιχθεί πάρα πολύ ε, ή εξελιχθεί ως άνθρωποι σε ό,τι αφορά τη διοντολογία και την ηθική μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό και ενδεικτικό. Εμείς έχουμε ενώπιον μας λοιπόν ένα τεράστιο έργο και καθήκον έτσι ώστε να δοθούν κίνητρα και παροτρύνσεις ε, δια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλω να επισημάνω το εξής. Όσο υπάρχει ε, θεωρία για την επικράτηση ενός είδους ή την κυριαρχία θα υπάρχει και σεξισμός. Χρειαζόμαστε μια νέα ιδεολογία, μια νέα κουλτούρα ανοχής, καλοσύνης, ανθρωπιάς απέναντι σε όλους και δεν βοηθάει να έχουμε τέτοιες οργανώσεις ε, ανθρωπιστικές και να τους εκπαιδεύουμε πώς να συμπεριφέρονται σε γυναίκες σε περιόδους και περιοχές κρίσης. Δεν αρκεί αυτό. Θα πρέπει από την παιδική ηλικία εξαπαλώνων ήχων να μαθαίνει κανείς στην κοινωνία μας πώς συμπεριφέρεται στον άλλον. Και ο άλλος μπορεί να είναι άνθρωπος, μπορεί να είναι όμως και ζώο. Ευχαριστώ πολύ. Muchas gracias, Σας ευχαριστούμε κύριε Χαίπ. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση για το σημείο αυτό και περνάμε στο επόμενο, το σημείο 17, με θέμα τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων. Θα ακούσουμε την παρουσίαση μιας μελέτης που έγινε από το Τμήμα Πολιτικών και έχει αντικείμενο τη συνεκτίμηση του φύλου στον κοινοτικό προϋπολογισμό και γενικώ τη συνεκτίμηση του φύλου στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Το συζητούμε εδώ και πολύ καιρό και χαίρομαι για την ευκαιρία που έχουμε να ακούσουμε την παρουσίαση αυτής της μελέτης που θα την αξιοποιήσουμε και στη συνέχεια στις εκθέσεις μας αλλά μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η πτυχή του προϋπολογισμού και το πώς συμπεριλαμβάνεται η ισότητα των φύλων σε αυτό. Παρακαλώ τους καλεσμένους μας να έρθουν στο Προεδρείο για να μας κάνουν την παρουσίαση. Muy bien, pues eh, para... Ωραία. Αρχίζει. Λοιπόν, η παρουσίαση, ε, η κυρία Μαργαρίτα Σάνς πρώτη θα λάβει το λόγο για να μας εισαγάγει στο θέμα, αν είναι έτοιμα όλα τα τεχνικά ζητήματα. Thank you very much, Chair. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ για την πρόσκληση να παρουσιάσουμε αυτή τη μελέτη για τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ισότητα των φύλων. Η Επιτροπή Γυναικών ζήτησε από την Πλόμε και Sands να κάνουμε αυτή τη μελέτη από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο του 2015 πώ έχει γίνει η έρευνα με δευτερογενή στατιστική ανάλυση, desk research και ε, συνεντεύξεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλου. Ε, από την Αυστρία, Σουηδία και Γερμανία ενεχομένως. Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω, να σας συστήσω τους εμπειρογνώμονές μας. Έχουμε την καθηγήτρια κυρία Φιώνα Μπέβεριτς και την δόκτωρα ε, ε, Φιράτ Τσενγκής από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ. Η κυρία Φιώνα Μπέβεριτς είναι Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ στο τμήμα κοινωνικών επιστημών και ασχολείται ιδιαίτερα και ειδικεύεται στην ισότητα των φύλων. Έχει ιδιαίτερη ε, εμπειρία στην συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου και πώς εφαρμόζεται στις πολιτικές ε, των διεθνών οργανισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Η κυρία Φύρα ε, Τσέγγις είναι στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ στη νομική σχολή έχει λάβει υποτροφία Marie Curie και ασχολείται με την οικονομική διακυβέρνηση, ε, σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και ισότητα φίλων και είναι ε, λέκτορας. Θα, της δώσω, θα δώσω το πρώτο το λόγο στη Φιώνα. Σας ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σας. So our task, our task was Ο στόχος μας ποιος ήταν να δούμε αν μπορούμε να βρούμε μια μεθοδολογία για να χρησιμοποιήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς μπορεί να γίνει ένας προϋπολογισμός με βάση το φύλλο, πώς να βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλους ενεχομένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να είναι πιο αποτελεσματική. Έχουμε εντοπίσει τρεις πιθανούς δυνατούς τρόπους για να βοηθήσει ενδεχομένως ε, αυτό ε, στην εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον προπολογισμό πάντα μιλώντας. Ε, πρώτη πιθανή χρήση είναι να ελέγχουμε συστηματικά και τακτικά τον προπολογισμό για να δούμε κατά πόσο η ε, δεσμεύσει υψηλού επίπεδου για την ισότητα των φύλων βρίσκουν ανταπόκριση στον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα κονδύλια. Δηλαδή είναι ένας τρόπος, αν παρακολουθείς που πηγαίνουν τα χρήματα, να διαπιστώνεις εάν αυτή η δέσμευση που έχει αναλυφθεί σε υψηλό επίπεδο μεταφράζεται στην καθημερινή πρακτική ε, στη ροή των κονδύλιων. Δεύτερον, για ποιο λόγο είναι αποτελεσματική εφόσον είναι ε, ε, αυτή η τακτική είναι ακριβώς επειδή συνεκτιμάται το φύλλο σε όλες τις πολιτικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί σε ε, υψηλό επίπεδο και θα πρέπει να αντανακλάται αυτό και στην καθημερινή εκτέλεση του προπολογισμού. Τρίτος τρόπος είναι να εξετάζουμε το προπολογισμό και να βλέπουμε εάν προωθείται η ισότητα και να υπάρχει ένα σύστημα αναφοράς για το αν προχωρούμε προς την ισότητα των φύλων και αυτό μπορεί να οδηγεί σε αναθεώρηση και ανασχεδιασμό των πολιτικών και των στρατηγικών. Δηλαδή, ο προπολογισμό είναι μια ευκαιρία παρέμβασης, είναι ένα εργαλείο για διάφορους φορείς συμπεριλαμβανομένου και του Κοινοβουλίου να μπορέσουν να μετρούν την πρόοδο και να την αξιολογούν. Αυτά λοιπόν τα τρία μαζί μας κάνουν να θεωρούμε ότι ο προϋπολογισμός μπορεί να θεωρηθεί εργαλείο διακυβέρνησης, οικονομικής και πρόθεσης της δημοκρατικής νομιμότητας. Θα σας εξηγήσουμε τη μεθοδολογία μας και θα σας πούμε πώς την εφαρμόσαμε, το βλέπετε κι εσείς και στο τέλος θα υποβάλουμε κάποια ερωτήματα για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτή η μεθοδολογία στην πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Τσέγγις. Χαίρομαι που βρίσκομαι ενώπιό σας να σας δώσω μια βασική ενημέρωση για τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε, πώς την αναπτύξαμε και πώς μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τη συμπεριλάβει ε, στη δική του προσέγγιση για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να αποφασίζει στο μέλλον ή αποφασίσει ότι θα έχει μια ε, προσέγγιση ισότητας και φύλου γενικότερα στον προπολογισμό. Στην έκθεση αυτή παρουσιάζουμε μια γερή, στιβαρή μεθοδολογία ενδεχομένω που θα δημιουργήσει τη δυνατότητα να έχουμε ένα εξωτερικό ορόσημο, ε, benchmark, για να δούμε όχι πώς λειτουργούν οι πολιτικές, αλλά πώς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αν θέλουμε να τις βελτιώσουμε ως προς την ισότητα φύλου. εσκεμένα έχουμε υιοθετήσει αυτή την προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή και θα βρείτε αναλυτικά στοιχεία στο παράρτημα υπαριθμών 1. Ε, το βασικό στοιχείο είναι ότι μια δημοκρατική προσέγγιση ε, παροχής δυνατοτήτων θα πρέπει να είναι ένα δημοκρατικό εργαλείο δημοκρατικής διακυβέρνησης και δεν αρχίζουμε λοιπόν από τα χρήματα, εμείς δεν σκεφτόμαστε αριθμούς, έχουμε ξεπεράσει αυτές τις λογικές, κοιτούμε τι δυνατότητες θα πρέπει να έχουν οι άνθρωποι και τι πρόσβαση αν θέλουν να ζουν μια ζωή αξιοπρεπή, πλήρη και ολοκληρωμένη. Από εκεί ξεκινάμε και όχι από τα χρήματα. Δεύτερον, επιλέγουμε ε, κάποιους τίτλους του προπολογισμού για να δούμε ε, πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτή η μέθοδος σε περίπτωση που αποφασίσει το Κοινοβούλιο στο μέλλον να υιοθετήσει αυτή την προσέγγιση γενικά στον προπολογισμό. Κάτι που θα τονίσει και πάλι στο τέλος η Φιώνα. Τονίζουμε ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει τεράστιο χάσμα δεδομένων για το ε, ε, πώς αξιολογείται από πλευρά ισότητας φύλου η κάθε δαπάνη του προϋπολογισμού. Και αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και να έχουμε αυτή την προσέγγιση με βάση το φύλο, χρειαζόμαστε πολλά περισσότερα συστηματικά δεδομένα που να συλλέγονται συστηματικά, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους και τους συμμετέχοντες στην κοινοτική χρηματοδότηση γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο τέλος, Βάσει των παρατηρήσεών μας έχουμε και κάποιες συστάσεις για προγράμματα σημεία δράσης των θεσμικών οργάνων αν θέλουν να βελτιώσουν την ισότητα φύλου στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά η διαδικασία του προπολογισμού ε, εμπλέκει και τα κοινοβούλια που ζητούν απόδοση λογαριασμών και Οπότε με τη συνεκτίμηση του φύλου στον προπολογισμό δεν θα βελτιωθεί μόνο η ισότητα των φύλων, αλλά και η οικονομική και η δημοκρατική λογοδοσία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ τα κοινοβούλια. Πριν αναφέρθηκα σε κάποιε ε, ικανότητες, πρόκειται κάποιε στοιχειώδει πληροφορίε, ε, Μπορεί να φαίνεται αόριστο αυτό το θέμα των ικανοτήτων. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα. Χρησιμοποιούμε πέντε ομάδες ε, και τις συνοψίζουμε στην μελέτη αυτή Μιλούμε ε, για την ανάμειξη των γυναικών στην κοινωνία, το ρόλο τους στις οικογενειακές δομές, στις αποφάσεις και σε άλλες ε, δομές ε, εξουσίας στην κοινωνία καθώς και την ένταξή τους στο, στο πολιτικό σύστημα, στην παιδεία, στην οικονομία και σε άλλες δομές εξουσίας. Επίσης, η δέσμευσή τους στράτευσή τους ως προς το περιβάλλον, το δικαίωμα στη στέγη και το δικαίωμα να ζουν σε μια αρμονική και ειρηνική συνύπαρξη με τα υπόλοιπα είδη και κατά πόσο μπορούν να εκπληρώσουν τα χόμπι τους, ε, να κάνουν τις ελεύθερες επιλογές τους, αν έχουν ελεύθερο χρόνο και επίσης ε, ανάμεξη, ε, αντέσμευση ανδρών και γυναικών, ε, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την ηλική διάσταση του σώματός τους, αλλά και την συναισθηματική πτυχή του σώματος. Σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία, πέντε βήματα ακολουθήσαμε. Σας μίλησα για τις ικανότητες που και στη βιβλιογραφία θεωρούνται βασικός παράγοντας για την διαβίωση ανδρών και γυναικών και την ανάμειξή τους στις ε, κοινωνικές δομές και στις δομές εξουσίας. Οπότε το πρώτο βήμα είναι εντοπισμός και αναγνώριση αυτών των ικανοτήτων. Δεύτερο βήμα τη συντεριάξαμε με τις διάφορες πολιτικές που καλύπτονται από το κοινοτικό προπολογισμό για να δούμε σε ποιο βαθμό τα δημοσιονομικά κονδύλια ή συγκεκριμένες δημοσιονομικές γραμμές μπορούν να επηρεάσουν συγκεκριμένα την ισότητα των φύλων. Τρίτο βήμα, ανάλυση των ε, στόχων της πολιτικής κάθε δημοσιονομικής γραμμής για να δούμε αν η πιθανή συνέπεια στην ισότητα φύλων αναγνωρίζεται και λαμβάνεται υπόψη στη δημοσιονομική διαδικασία. Επίσης ε, εξετάζουμε τα στοιχεία, τα δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να δούμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι του κοινοτικού προϋπολογισμού σε κάθε δημοσιονομική γραμμή και ανάλογα με τη γενική επισκόπηση που κάνουμε και την εικόνα που δημιουργούμε υποβάλλουμε κάποιες σκέψεις ε, και κάποιες συστάσεις για αλλαγές ε, στις πολιτικές. Και μάλιστα έχουμε και μια σύνοψη των πορισμάτων μας για να λυθούν πιο εύκολα υπόψη και να γίνουν πιο ευανάγνωστοι και κατανοητά εξηγούμε τι σημαίνει κάθε τμήμα του πίνακα. Για παράδειγμα, ε, το Ταμείο ε, παροχή Βοήθειας προς Απόρους. Στόχος είναι να στηριχθούν οι κοινωτικές δράσεις και να δοθούν ε, να δοθεί αρρωγή στους πλέον απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε αντίστοιχη κατηγορία στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Έτσι μπορούμε να εντοπίσουμε τους στόχους πολιτικής του συγκεκριμένου κεφαλαίου Επίσης βλέπω το φάσμα της ισότητας των φύλων και τις συνέπειες ε, του συγκεκριμένου κεφαλαίου στην ισότητα των φύλων. Όταν μιλούμε για φάσμα βλέπουμε τι μπορεί, ε, που μπορεί να επηρεάσει το συγκεκριμένο δημοσιονομικό κεφάλαιο. Και σε ό,τι αφορά τις συνέπειες στην ισότητα των φύλων, βλέπουμε αν οι συνέπειες αυτές, αν ο αντίκτυπος αυτός είναι άμεσος ή έμεσος ή μικρός, μεσαίος ή μεγάλος. Επίσης, ε, Είχαμε και εμπειρική και θεωρητική εξέταση της ε, βιβλιογραφίας για να δούμε ποιοι είναι οι διαρθρωτικοί λόγοι και τα αίτια της ανισότητας στις συγκεκριμένες τομείς. Βλέπουμε την κατανομή των κεφαλαίων και αναζητούμε ε, κοινοτικά δεδομένα σε ό,τι αφορά τους ε, δικαιούχους συγκεκριμένου κεφαλαίου. Στη μελέτη αυτή εξετάσαμε έξι διαφορετικά κεφάλαια του προϋπολογισμού. Βέβαια, επειδή είχαμε περιορισμό και χώρου και χρόνου, σκεφτήκαμε ότι είναι σημαντικό να αντιληφθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι αν η συνεκτίμηση του φύλου στον προπολογισμό χρησιμοποιηθεί ω εργαλείο, θα πρέπει να καλύπτονται όλα τα κεφάλαια του προπολογισμού, γιατί όλε οι πολιτικέ έχουν κάποιο αντίκτυπο στην ισότητα των φύλων. Αν και μερικέ φορέ ε, είναι πιο συγκαλυμμένο και έμεσο αυτό ο αντίκτυπο. Όπως είπα και στην αρχή, όταν μίλησα για τις ικανότητες, θα πρέπει να ξεπεράσουμε τους αριθμούς. Ο κοινοτικός προϋπολογισμός είναι σχετικά χαμηλός σε σχέση με τους εθνικούς. Βέβαια, εδώ το μέγεθος ε, δεν ενδιαφέρει. Και μέσω των κινήτρων που δίνουμε σε εθνικό επίπεδο για τις ε, αποφάσεις των δαπανών, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός ε, καλύπτει σημαντικά κενά εκεί που ιστερεί η κρατική συμμετοχή. Έχουμε μερικά παραδείγματα θετικά και αρνητικά, όπου βλέπουμε πόσο δυνάμει, ο δυνητικός κίνδυνος της, των ευρωπαϊκών δαπανών ε, είναι μεγάλος. Επίσης, ε, έχουμε τον ορίζοντα 2020 και το πώς επηρεάζει την ισότητα των φύλων. Το ακούσαμε και στην προηγούμενη έκθεση οι στόχοι ισότητας των φύλων του ορίζοντα 2020 δυστυχώς δεν υλοποιούνται. Σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον. Σε σχέση όμως με άλλα κεφάλαια, βλέπουμε ότι το ορίζοντας 2020 και η έρευνα και η επιστήμη είναι από, τους πιο, από τα πιο σημαντικά κεφάλαια του προπολογισμού που περιλαμβάνουν κριτήρια ισότητας φύλου και για την επιλογή της χρηματοδότησης και για την ε, σύνθεση των ε, επιστημονικών και τεχνικών πάνελ. Οπότε στην πράξη, για την εφαρμογή του προγράμματος Horizon 2020, αυτό αφορά περισσότερο για τους μελλοντικούς ε, ερευνητές που ευελπιστούμε ότι θα φέρουν μια άλλη προοπτική για την μελλοντική κατεύθυνση των πόρων και των προγραμμάτων. Και προετοιμάζουμε σήμερα τις γυναίκες ερευνητές για πιο σημαίνοντε ε, και ηγετικού ρόλου στο μέλλον σε θέματα έρευνα. Σε ό,τι αφορά τι βιομηχανικέ σχέσει και τον κοινωνικό διάλογο, δεν έχουμε σημαντική δέσμευση υπέρ τη ισότητα των φύλων. Ενώ θέλουμε να είναι ισχυρή η παρουσία και των ανδρών και των γυναικών στη διαμόρφωση του προγράμματο Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμω ήταν ένα αρνητικό πόρισμα από την ανάλυση του προπολογισμού και για, το, για το Creative Europe για την ε, Δημιουργική Ευρηματική Ευρώπη, το κεφάλαιο 1504. Εκεί υπάρχει μια διαρθρωτική ανισότητα και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ευκαιρία εκεί να βελτιώσει την ισότητα των φύλων με την θέσπιση κριτηρίων για την κατανομή των κονδυλίων. Δυστυχώς όμως δεν ε, αξιοποιήθηκε αυτό το δυναμικό στον προϋπολογισμό. Και να ξαναδώσω το λόγο στη Φιώνα αφού σας ανέλησε τη μεθοδολογία μας. Ευχαριστώ. Έχουμε τρία βασικά ευρήματα από την ε, μελέτη. Το πρώτο είναι ότι η δέσμευση για την ισότητα των φύλων δεν ε, ακολουθείται από ικανές δαπάνες. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα θέμα ιδιαίτερα προβληματικό. Όταν τα θέματα της ισότητας των φύλων ε, δεν αντιμετωπίζουν ε, κατάλληλα, διότι υπάρχει μια εγκάρσια σχέση. Το δεύτερο έρημα είναι ότι οι τίτλοι του προπολογισμού δεν είναι πάντα διάφανοι και δεν εφαρμόζεται, ε, κατά πόσο μάλλον εφαρμόζεται το mainstreaming στον προπολογισμό. Και το τρίτο έβριμα, αυτό αφορά το χάσμα μεταξύ των ε, φύλων, ότι δεν υπάρχουν κατάλληλα <clears throat> στοιχεία και δεδομένα τα οποία συχνά ούτε καν συλλέγονται. Όπως είπα νωρίτερα, σχέση με τον ορίζοντα 2020 δεν υπάρχει μηχανισμός για να επανεξεταστεί το ζήτημα και να αλλάξουν τα κριτήρια και βασιζόμαστε σε εξωτερικές μελέτες Λοιπόν, οι συστάσει μα πρώτα ότι η ισότητα των φύλων θα πρέπει να αναγνωριστεί ω στόχος πολιτική σε όλου του τίτλου προπολισμού, Δεύτερον, το gender mainstreaming θα πρέπει να ε, εφαρμοστεί στην πολιτική σε όλους τους τίτλους σε όλα τα κεφάλαια του προπολισμού. Τρίτον, τα ε, στοιχεία τα οποία ε, δίνονται από τον προπολογισμό θα πρέπει να διευκρινιστούν και να αυξηθεί η διαφάνεια τρίτον, τα... οι δείκτες σχετικά με τον φύλλο θα πρέπει να αναπτυχθούν συστηματικά και να δημοσιευθούν. Δίχως αυτά τα τέσσερα στοιχεία που προανέφερα δεν μπορεί να είναι πραγματικά ουσιαστική η υλοποίηση του προπολογισμού. Τώρα, τα θεσμικά όργανα και τα υπηρεσίες της ε, Ένωσης θα πρέπει να χρησιμοποιούν την ε, δείκτες η Κομισιόν θα έχει ένα διαρματίσει σημαντικό ρόλο για την εφαρμογή αυτών των συστάσεων και ότι ο προπολογισμό θα είναι επαρκώς διαφανής. Το Ευρωγενοβούλιο έχει να διαρματίσει σημαντικό ρόλο για την έγκριση και την απαλλαγή. Σας θέτω τώρα κάποιες ε, κάποια ερωτήματα κατά πόσο χρήσιμη είναι η μεθοδολογία μας σχετικά με τον εντοπισμό αδυναμιών στον πολιτική για την ισότητα των φύλων. Κατά πόσο το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι αυτές οι προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με την έλλειψη σαφών δεδομένων. Θα μπορούσε να προσθέσει το, αυτή η διαδικασία μεγαλύτερη αξία στις εργασίες της, του Κοινοβουλίου. Και κατά πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το, αυτή η συνεκτίμηση του φίλου του προπολογισμού για τις δολοτικές εργασίες τώρα. Το λόγο έχουν οι συνάδελφοι, αλλά έχουμε μόνο τρία λεπτά στη διάθεσή μας Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτή η έννοια του gender budgeting. Χρειάζεται καταρχήν να ε, εστιάσουμε στους ε, σημαντικούς προϋπολογισμούς. Δεν θα θέλαμε να ε, ασχοληθούμε με τους μικρούς προϋπολογισμούς. Εγώ θα ήθελα να θίξω το θέμα του αγροτικού προϋπολογισμού με τις άμεσες πληρωμές, άμεσες ενισχύσεις. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τι γίνεται πίσω από αυτές. Εάν αυτές οι εκμεταλλεύσεις οι οποίες λαμβάνουν τα κονδύλια διευθύνονται από άνδρες, μόνο να γνωρίζουμε ότι και γυναίκες εργάζονται στο τομέα της γεωργίας. Θα πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης αυτής της εκμετάλλευσης. Είναι ένα ζευγάρι ή αποκλειστικά ο άντρας, ο σύζυγος. Όλα αυτά είναι στοιχεία ιδιαίτερα σημαντικά, διότι οι άμεσες επιδοτήσεις στον γεωργικό τομέα, άμεσες ενισχύσεις στον αγροτικό τομέα αποτελούν το πιο σημαντικό τμήμα των αγροτικών δαπανών. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι γίνονται οι επιχειρήσεις, ε, αν είναι ε, αμυγός ε, ανδροκρατούμενες ή όχι. Έχει σημασία πού πηγαίνουν τα κονδύλια. Θα μας απασχολήσει λοιπόν πολλά χρόνια ακόμα αυτό για να δούμε πού πηγαίνουν τα χρήματα. Το επόμενο βήμα να κανονίζουμε να φτάνουν σε καλύτερα χέρια ή σε χέρια γυναικεία ε, είναι πολύ μακρινό γιατί βλέπουμε ότι ε, όταν ρωτάμε εμεί οι βουλευτές που πηγαίνουν τα χρήματα είναι ε, αποσπασματική η πληροφόρηση για τον τελικό δικαιούχο διότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία και δεδομένα για τα χρήματα που έρχονται για την προστασία του περιβάλλοντος, τα κοινωνικά, τα γεωργικά, τα διαρθρωτικά ε, όλα αυτά τα κονδύλια δεν τα ξέρουμε και, γιατί υπάρχουν και ε, πολλά κονδύλια από τη συγχρηματοδότηση με συμμετοχή των κρατών μελών. Και πώς τελικά με τη συγχρηματοδότηση αυτά τα χρήματα ε, παρεκτρέπονται, πώς να το πω, και καταλήγουν σε ανδρικά χέρια, ενώ κανονικά πρέπει να είναι ουδέτερας προς το φύλλο. Δεν ξέρω, θέλετε να προσθέσετε τίποτα. Συμφωνώ ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σε όλη τη διάρκεια της δημοσιονομικής διαδικασίας τέτοια δεδομένα, γιατί μας οδηγεί στα κράτη-μέλη και στη χρηματοδότηση. Χωρίς τέτοια στοιχεία δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν υπονομεύεται η ισότητα του φύλου ή ενισχύεται. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Η κοινή γεωργική πολιτική είναι ένας από τους τομείς μαζί με την περιβαλλοντική πολιτική που επισημάναμε ιδιαίτερα και αναδείξαμε στη μελέτη και πολύ σημαντικός κλάδος και για το μέλλον. Και γίνονται κάποιες εμπειρικές μελέτες, ε, στην Ιρλανδία συγκεκριμένα, σε επιμέρους τομείς, αλλά συμφωνώ και με σας και με τη Φιώνα ότι πολύ δρόμο έχουμε ακόμη μπροστά μας, γιατί χρειαζόμαστε αξιόπιστα και ακριβή στοιχεία για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα πορίσματα. Σας ευχαριστώ θερμά ε, για τη μελέτη που μας παρουσιάσετε. Ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο της ημερήσης διάταξης και περνάμε στο τελευταίο, το μισθολογικό, ή μάλλον το συνταξιδοτικό χάσμα και τις ηλικιωμένες γυναίκες που διαβιώνουν μόνες τους. Ε, ενημέρωση για τις συνθήκες διαβίωσης τους. Παρακαλώ τους εμπειρογνώμονές μας να μας κάνουν την εισαγωγή. Um, hi again, everybody. Um, I'm actually here to present. Ευχαριστώ. Να σας παρουσιάσω δύο μελέτες που έχουν γίνει σε αυτό τον ε, σημαντικό τομέα Μπορείτε να δείτε αναφορά στις δύο μελέτες σε αυτή την διαφάνεια. Νομίζω πως δεν χρειάζεται να υπογραμμίσω πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια σαφή εικόνα πως ακόμα και στην συνταξιοδότηση υπάρχουν τεράστιες διαφορές εισοδημάτων ανάμεσα στους άντρες και γυναίκες διότι μέχρι τώρα είχαμε επικεντρωθεί μόνο στην αγορά εργασία Ορισμένοι από εσά <clears throat> ίσως να έχετε δει κάποιε από αυτές τις μελέτες, αλλά θα θέλω να δώσω κάποιε παραπάνω λεπτομέρειες και προφορίες. Γιατί είναι σημαντικό πρώτα απ' όλα. γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές μεταξύ άνδρων και γυναικών. Είναι ζήτημα ισότητας, ζήτημα ανεξαρτησίας και είναι θέμα φτώχειας. Τώρα, η φτώχεια ίσως έχει τονιστεί ιδιαιτέρως, έχει σημασία για το χάσμα μεταξύ των ανδρών και γυναικών σε ό,τι φορά τη σύνταξη. Αλλά ποιο είναι το ζήτημα. Ο λόγος που υπάρχει αυτό το χάσμα, αυτό που παίζει σημαντικό ρόλο εδώ είναι η ανεξαρτησία και η ισότητα. Μπορούμε να επανέλθουμε στην προηγούμενη διαφάνεια και μετά να ξαναπροχωρήσουμε στην άλλη. Αυτό με κάποιο τρόπο εξηγεί την σειρά των που έχει ακολουθηθεί από τις μελέτες. Ε. Εδώ η πρώτη έγινε το 2013 και μπορείτε να την βρείτε στο διαδίκτυο. Η άλλη θα εμφανιστεί στο διάκτυο σύντομα τον Ιούνιο και θα μπορείτε να την βρείτε και στο διαδίκτυο. Την έχει αναλάβει η... το τμήμα ισότητας του Ειδική Διεύθυνση δικαιοσύνη. και θα έλεγα ότι εστιάζουμε σε δύο διαφορετικές ε, ηλικιακές ομάδες η πρώτη αφορά τους ηλικιωμένους γενικότερα και από στατιστική σκοπιά, όπως γνωρίζετε, ορίζουμε ως ηλικιωμένους τους, τα πρόσωπα που είναι άνω των 65. Η δεύτερη μελέτη δεν επικεντρώνεται στους ηλικιωμένους αλλά στην ομάδα που μπορείτε να ορίσετε ως ε, νεαρούς ηλικιωμένους, νεότερους ηλικιωμένους. Ας δούμε λοιπόν τους ε, πολιτικές αιτίες ε, για τους οποίους η Κομισιόν ενδιαφέρονται για αυτά τα φαινόμενα διότι μπορούν να οδηγήσουν σε ε, εφαρμογή πιο καλύτερων, πιο καλών πολιτικών. Εάν εστιάσουμε στους νέους, νεότερους ηλικιωμένους θα πρέπει να δούμε ότι τα στοιχεία αφορούν αυτά τα πρόσωπα. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που εν μέρης συνδέεται με την ανεξαρτησία και είναι το εξή. Εάν εστιάσετε στους ηλικιωμένους, τους ιδιαίτερα ηλικιωμένους, δηλαδή 80 και πλέον ετών, τότε το χάσμα μπορεί να είναι χαμηλότερο διότι υπάρχουν ε, τα ε, παράγωγα δικαιώματα και αυτό λόγω των, ε, του θέματος ότι υπάρχουν ε, ε επιζήσεις, επιβιώνοντες, ε, κάποιοι που έχουν επιβιώσει περισσότερο. Αυτά, αυτό είναι ο λόγος για τους οποίους οι δύο διαφορετικές εκθέσεις αφορούν, μελέτες αφορούν δύο διαφορετικά ηλικιακά όρια. Αυτή θα πρέπει λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά και στις δύο ομάδες όταν περάσουμε τώρα στην επόμενη διαφάνεια καταρχήν τι ακριβώς ε, μετρούμε μετρούμε δύο πράγματα υπάρχουν δύο βασικοί δείκτες ο πρώτος είναι πως τα άτομα εισπράττουν πόσοι μάλλον εισπράττουν συντάξεις Αυτό είναι ένας πρώτος δείκτης και ποια είναι η διαφορά μεταξύ άνθρωπων και γυναικών σε αυτόν τον δείκτη και το δεύτερο θέμα είναι ποια είναι η ποσοστία διαφορά στις ε, μέσων νέων των συντάξεων που οι γυναίκες λαμβάνουν σε σχέση με το μέσο όρο των ανδρών, των συντάξεων των ανδρών. Επανερχόμαστε τώρα στην προηγούμενη διαφάνεια. Όπως βλέπετε, οι δύο πρώτες ε, αριστερά μετρούν το χάσμα και η διαφορά είναι 40 έως 38% γύρω στο 40% και το δεύτερο είναι οι κολόνες ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες όπου αυτή η διαφορά είναι πιο περιορισμένη και είναι της του 5 με 6%. Πού είναι το πρόβλημα λοιπόν? Το χάσμα στο συνταξιοδοτικό, δηλαδή μεγάλες διαφορές μεταξύ των συντάξεων, μεταξύ των, των γυναικών και των ανδρών, σε ό,τι αφορά τη μέση σύνταξη. 40% υψηλό ποσοστό και μπορεί να μην ανταποκρίνεται στις δικές σας γνώσεις για την αγορά εργασίας, γιατί ο βασικός δείκτης δείχνει την ε, βασική διαφορά, τη μέση διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών στους μισθούς, τη μισθολογική ε, μέση διαφορά. Οπότε το στοιχείο που έχετε στο μυαλό σας για τη διαφορά είναι γύρω στο 16%. Τεράστια διαφορά λοιπόν μεταξύ των δύο ποσοστών μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος. Γιατί? Γιατί το μισθολογικό χάσμα του 16%, αυτό είναι ο κοινοτικός μέσος όρος εννοείται, δεν λαμβάνει υπόψη πολύ σημαντικές διαφορές που υπάρχουν στις ικανότητες των γυναικών ε, να βγάλουν ε, χρήματα. Αυτό το 16%, αυτή η διαφορά το 16% καταμετρά τις διαφορές ε, στο, στο, στο μισθό ανά ώρα. Αλλά οι γυναίκες εργάζονται πολύ λιγότερες ώρες σε σχέση με τους άνδρες. Οπότε αν λάβουμε υπόψη και αυτές τις διαφορές, καταλήγουμε το ίδιο περίπου ποσοστό με αυτό του συνταξιοδοτικού χάσματος, το 40% δηλαδή. Εδώ βλέπουμε δύο στήλε. Η μία έχει το συνταξιοδοτικό εισόδημα και το χάσμα στο συνταξιοδοτικό εισόδημα και η δεύτερη στήλη είναι μία νέα στατιστική πληροφορία που, έχει, που παρουσιάζει το συνολικό χάσμα στα εισοδήματα. Ποιο είναι το συνολικό χάσμα των εισοδημάτων. Αν πάρουμε τη μέση γυναίκα και τον ε, σε ηλικία εργάσιμη. Γιατί μια γυναίκα μπορεί να εργάζεται λιγότερες ώρες από έναν άντρα. Πολύ συχνά επίσης αμείβεται λιγότερο από έναν άντρα. Οπότε, αν τα λάβουμε υπόψη και αυτά, να λάβουμε υπόψη και αυτές τις διαφορές. Τις διαφορές των αριθμό ωρών, στη συμμετοχή της απασχόλησης, τότε καταλήγουμε σε ένα μέσο όρο που αγγίζει το 40% στις διαφορές ε, των εισοδημάτων. Οπότε το μήνυμα είναι το ότι ουσιαστικά το χάσμα στις συντάξεις αντικατοπτρίζει πλήρως ε, το μισθολογικό χάσμα, το χάσμα στα εισοδήματα. Και οι χαμηλές συντάξεις αντανακλούν ε, τις χαμηλές αμαρδές και τη λιγότερη απασχόληση των γυναικών. Είναι λογικό, οι γυναίκε δουλεύουν λιγότερε ώρε και ε, αμείβονται λιγότερο, να έχουν τελικά και χαμηλότερε χαμηλότερες Εδώ θα βάλω τέλεια. Με ένα ακόμη σχόλιο όμως. Φυσικά υπάρχουν μεγάλες διαφορές αυτό το 40% μεταξύ των χωρών. Δεν ισχύει το 40% για όλες τις χώρες. Σε μερικές χώρες το χάσμα είναι ε, μικρότερο και σε άλλες μεγαλύτερο. Τώρα, ε, πού οφείλεται το μικρό χάσμα όταν οι διαφορές είναι μεγάλες στην αγορά εργασίας. Αυτό οφείλεται στην, ε, στην πολιτική. Εξού και η ανάγκη συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων. Αυτά όμως θα σας τα πει η Εμμανουέλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν έχουμε χρόνο. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα, αλλά θα επανέλθουμε οπωσδήποτε. Τώρα θα δώσω το λόγο στη Μανουέλα Σάμακ και μου λέγουν ότι οι διερμηνείς θα μείνουν πέντε λεπτά παραπάνω κοντά μας. Έχουμε ένα δεκάλεπτο περίπου. Ε, ευχαριστώ. Ε, η εστίαση ε, ε, αυτού, του θέματος είναι για γυναίκες ηλικιωμένες που ζουν μόνες τους. Είναι μια ενημέρωση μιας πολύ παλιά μελέτης και προσπαθούμε να δούμε τι ζουν οι γυναίκες αυτές, ιδιαίτερα ηλικιωμένες που ζουν μόνες τους και κλείνει το μικρόφωνο της ομιλήτρης. Ε, ποιες αλλαγές έχουμε στις ε, συνταξιοδότηση, στις συντάξεις και στην ενεργό και πώς επιδρά η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στις γυναίκες εκείνες που ζουν μόνες τους. Target, it is... Ε, γιατί έχει σημασία Οι ηλικιωμένε ε, αυξάνονται σε αριθμό ιδιαίτερα στους ζουν μόνες τους για λόγους δημογραφικούς αλλά και για λόγους κοινωνικών αλλαγών στις οικογενειακές ε, δομές και ε, συγκρότηση. Το 2014 οι γυναίκες άνω των 65 ετών που ζουν μόνες τους στα 28 κράτη-μέλη ήταν περίπου 20 εκατομμύρια. 20 εκατομμύρια, δηλαδή 8% του γυναικείου πληθυσμού. Πολύ περισσότερο από άνδρες ηλικιωμένου που ζουν μόνοι τους, που είναι 7 εκατομμύρια, μόλις 3%. Ε, in the younger... Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι ε, στις... Ε, Μικρότερε ηλικίε ε, ε, του εργασιακού βίου, οι άντρε που εργάζονται και ζουν μόνοι τους, ε, είναι περισσότεροι από τις γυναίκες που ζουν μόνες τους. Όσο περνάει η ηλικία, αλλάζει αυτό. Θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν πώς επηρεάζει αυτή την ομάδα γυναικών η κάθε αλλαγή στα συστήματα των συντάξεων και στι μεταρρυθμίσει αυτέ. Να δούμε ένα δείκτη λοιπόν που έχει να κάνει με τον κίνδυνο φτώχειας και τις δυσκολίες να τα βγάζουν πέρα. Τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας και τα δεδομένα μας δείχνουν ότι οι ηλικιωμένε που ζουν μόνες τους ε, κινδυνεύουν πολύ περισσότερο να πέσουν στη φτώχεια κατά μέσο όρο από ότι οι άνδρες που ζουν μόνοι τους ή από γυναίκες που ζουν με άλλα πρόσωπα. Δηλαδή δεν είναι ανεξάρτητες οικονομικά οι γυναίκες αυτές που ζουν με άλλους αλλά δεν κινδυνεύουν να ε, ε, πέσουν και στην ένδυα. Μία στις τέσσερις ηλικιωμένε που ζουν μόνες τους έχουν ζητήματα φτώχειας να αντιμετωπίσουν σε σύγκριση με 19% ε, ηλικιωμένων ανδρών και μόνο 12% ε, είναι οι γυναίκες που δεν, οι ηλικιωμένες που δεν ζουν μόνες τους και είναι στη φτώχεια. Δεν θα σας ε, αναλύσω όλα αυτά τα στοιχεία, απλώς να σας πω το εξής που έχει σημασία. Όταν σκεφτόμαστε τις μεταρρυθμίσεις της συντάξης και τις αλλαγές στα συστήματα. Κοιτάξτε πόσες ηλικιωμένε που ζουν μόνες τους δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Στις ε, βορειοευρωπαϊκές χώρες είναι το χαμηλότερο ποσοστό, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες μόνες ηλικιωμένες έχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες να τα βγάλουν πέρα. Και το ίδιο ισχύει και για άλλες κατηγορίες ηλικιωμένων γυναικών, καλά και ανδρών, που ζουν μόνοι τους. Έτσι έχει λοιπόν η κατάσταση ποια ήταν η τάση ε, στις μεταρρυθμίσεις ε, των συντάξεων μέχρι τώρα. Έχουμε δει και ακούσαμε και από τη Φραντσέσκα και την παρουσίασή της ότι ε, η μισθολογική ψαλίδα μεταφέρεται και στη σύνταξη. Γιατί οι συντάξει είναι μια ανάκλαση των όσων συμβαίνουν στην αγορά εργασίας. Και όταν οι γυναίκε είναι σε χειρότερη μοίρα όταν εργάζονται, αυτό σημαίνει ότι όταν βγουν και στη σύνταξη, αντίστοιχα θα τους ακολουθήσει αυτή η κατάσταση και θα έχουν χαμηλότερε συντάξει. Πρόσφατες συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις προσπαθούν βασικά να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών ταμείων και συστημάτων. Δηλαδή, έχουν αυξήσει τη σχέση των συνεισφορών, των ασφαλιστικών εισφορών κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου και των επιδομάτων σύνταξης. Έχουν μειώσει το ρόλο της δημόσιας σύνταξης και έχουν ανατρέξει περισσότερο σε ε, συστήματα αυτασφάλισης, επαγγελματικής ασφάλισης και ιδιωτικής κατά κύριο λόγο. Αυτά τα μέτρα λοιπόν έχουν επηρεάσει αρνητικά τις γυναίκες χειρότερα από τους άντρες διότι εργάζονται σε πιο επισφαλείς συνθήκες και αυτό ε, επηρεάζει σημαντικά και αρνητικά το εισόδημά τους από τη σύνταξη σε προηγμένη, προχωρημένη μάλλον ηλικία. Ποιο είναι το πρόβλημα. Ορισμένες χώρες έχουν συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος ε, φτώχειας στους ηλικιωμένους, στους συνταξιούχους και ιδιαίτερα στις γυναίκες και ορισμένα κράτη λοιπόν αφού το κατάλαβαν προσπαθούν να το επιλύσουν. Και τι έκαναν. Προσπάθησαν να διευρύνουν την συνταξιδοτική κάλυψη, να αυξήσουν ε, τα επίπεδα επιδομάτων και να βελτιώσουν ε, τη σχέση ε, της ιδιωτικής ασφάλισης και της επαγγελματικής για να υποστηρίξουν και πρόσβαση για νέες γυναίκες ε, ηλικιωμένες και νέους με μη συνήθεις μορφές εργασίας, συμβάσεις. Έχει δείξει η κρίση ότι οι ε, επαγγελματικές συντάξεις και οι ιδιωτικές ε, συντάξεις ε, εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το τι συμβαίνει στην οικονομία. Λοιπόν, υπάρχει ένας κίνδυνος για τη βιωσιμότητα των ταμείων και των συστημάτων. οι συνέπειες αυτής της μεταρρύθμισης είναι γνωστές, τις είπαμε και προηγουμένως, όταν υπάρχει διαφορά με βάση το φύλλο στην ε, αγορά εργασίας στο μισθό, αυτό θα ενταθεί ακόμα περισσότερο στη σύνταξη. Και αυτό αυξάνει την εξάρτηση των γυναικών από το εισόδημα του συντρόφου τους. Το είδαμε από τα στοιχεία αυτά, ιδιαίτερα σε συστήματα πρόνοιας που βασίζονται σε σχέσεις και συντάξεις και δικαιώματα οικογενειακά περισσότερο από ατομικά όπως χώρες της Νότιας Ευρώπης ας πούμε. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι οι γυναίκες ζουν περισσότερο. Οπότε ζουν και ηλικιωμένες περισσότερο. Ε, οπότε, ε, όταν είναι χαμηλή η σύνταξή του υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος φτώχεια ιδιαίτερα για πάρα πολύ ηλικιωμένε, για υπερήλικες γυναίκε. Όχι αυτές που είναι τώρα υπερήλικες, αυτές που θα είναι αύριο υπερήλικες. Επίσης, το θέμα ε, των παράγωγων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα το τη σύνταξη επιζώντος. Σήμερα υπάρχει πολύ μεγάλη υποστήριξη ηλικιωμένων γυναικών που ζουν μόνες τους, ιδιαίτερα για τις γυναίκες που δεν έχουν ε, ιστορικό ε, εργασίας. Σε χώρες όπως είναι η Ιταλία ή άλλες χώρες της Μεσογείου, η ε, ψαλίδα η συνταξιοδοτική είναι πολύ μικρή γιατί οι ηλικιωμένες συχνά έχουν πρόσβαση ε, στη σύνταξη επιζώντος. Ε, αλλά όπως είπε και η Φραντσέσκα, από πλευράς οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών αυτό είναι πρόβλημα. Και ε, για γυναίκες που δεν έχουν παντρευτεί ποτέ είναι επίσης πρόβλημα, διότι δεν καλύπτονται από αυτά τα παράγωγα δικαιώματα της σύνταξη επιζώντος, αλλά έχουν συνεισφέρει με τη, τους φόρους τους και έχουν καταβάλει ε, εισφορές και σε πολλές χώρες ε, υπάρχει θέμα κινήτρου να εργαστούν οι γυναίκες αυτές. Ε, και γίνεται μια συζήτηση σε πολλές χώρες αν θα πρέπει να μειωθούν αυτά τα δικαιώματα και τα επιδόματα ε, και αντί να μειωθεί η φτώχεια για τις ηλικιωμένες που δεν έχουν δουλέψει πολύ στη ζωή τους να έχουμε ελάχιστη σύνταξη, ελάχιστο συνταξιωτικό επίδομα κατά κάποιο τρόπο. Ε, ένα ελάχιστο, ας πούμε, καθολικό εισόδημα του συνταξιούχου, πώς να το πω, για να μειωθούν οι αδικίες μεταξύ των γυναικών. Not going on this. Δεν θα επεκταθώ σε αυτό. Προσπαθώ να κλείσω για την πολιτική και τι συστάσεις θα δώσουμε. Το πρώτο ε, θέμα που έχει σημασία είναι για τις γυναίκες που είναι ανήπανδρες, ε, ανήπανδρες μητέρες, ε, νέες και λιγότερο νέες. Και γενικότερα γυναίκες που δεν, δεν παντρεύτηκαν ποτέ, που δεν ήταν ποτέ ε, ζευγάρι, δηλαδή που δεν μπορούν να υπολογίζουν στο εισόδημα του συντρόφου. Και το μεγάλο θέμα είναι να εισαχθούν με μονομένα ατομικά δικαιώματα κοινωνικά που δεν, εξαρτώνται, που δεν έχουν σχέση με συζυγικές ή οικογενειακές σχέσεις ή τον οικοκυριό. Δηλαδή θα πρέπει να εξετάζουμε ως μονάδα το άτομο και όχι την οικογένεια για να ε, μειωθούν αυτά τα αντικίνητρα προς εργασία και να υποστηριχθεί όλο αυτό το μερίδιο των γυναικών που ζουν μόνοι τους και αυξάνεται. Ε, ε, Λοιπόν, όλα αυτά τα ζητήματα είναι βασικά και γεγονωμένα και υπάρχουν και άλλα που έχουν σημασία όταν συζητούμε για τις συντάξεις. Women living alone. Ε, το πρώτο που είπα προηγουμένως είναι Use, uh, uh, universal... να χρησιμοποιήσουμε μια κατώτατη σύνταξη ενιαία καθολική που δεν έχει καμιά σχέση με το ιστορικό εργασίας του ατόμου, να υπάρχει ένα ελάχιστο εγγυημένο συνταξιδοτικό εισόδημα για γυναίκες που διέκοψαν ε, την καριέρα τους ή δεν είχαν ποτέ σταδιοδρομία παρά μόνο σύντομο εργασιακό βίο. Θα πρέπει να υποστηρίζεται πολύ περισσότερο η δεν ειχαν ποτε σταδιοδρομια παρα μονο συντομο εργασιακο βιο θα πρεπει να υποστηριζεται πολυ περισσοτερο πιστοση ε, για τη σύνταξη για περίοδους Ε, γονικής άδεια και ιδιαίτερα για τους άνδρες για την πατρική άδεια. Και επίσης να εθαρρύνουμε την μερική εργασία, τη μερική απασχόληση όταν ε, ε, μεγαλώνει κανείς τα παιδιά του και με ειδικά συστήματα απασχόλησης να προβλέπονται τέτοιου είδους διατάξεις. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά θα πρέπει να διακόψουμε θα μας φύγουν οι διερμηνείς. Ένα λεπτό για να ολοκληρώσετε. Στην έκθεση θα βρείτε και άλλες προτάσεις. Το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι με τα νέα συνταξιδοτικά συστήματα ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να υποστηριχθεί η εργασία και ο μισθός των γυναικών, σωστή αμοιβή όταν εργάζονται. Αλλιώς η σύνταξή τους κινδυνεύει να είναι πάρα πολύ χαμηλή και η εξάρτησή τους, συζυγική κτλ. θα τις οδηγήσει σε μεγάλα προβλήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση αυτή και τις δύο Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και πολύ θα θέλαμε να δώσουμε συνέχεια σε αυτό. Αν δούμε το ακροατήριο θα διαπιστώσουμε ότι οι περισσότερες είναι γυναίκες. Και μας ενδιαφέρει να μειώσουμε και την ψαλίδα αυτή και τη μισθολογική και τη συνταξιοδοτική. Ευχαριστώ πολύ. Λήξη της σημερινής συνεδρίασης. Επόμενη συνεδρίαση από τις 3 μέχρι τις 6.30 στις 30 Ιουνίου και ευχαριστούμε και τους διερμηνείς για την υπέρβαση ωραρίου. Iba posledná poznámka, ak sú nejaké otázky na obe if there are any questions, uh, you can address them to the secretariat. And, uh, Αν έχετε ερωτήσεις, να τα πείτε στη γραμματεία και με χαρά να απαντήσουν θα διαβαστούν γραπτό οι ερωτήσεις προς τις κυρίες που θα την παρουσίαση. επόμενη συνεδρίαση στις 13 Ιουλίου, λοιπόν, 3 με 6.30.